Uh, take your seats. I'm going to make... Καθίστε παρακαλώ, θα ξεκινήσω αμέσως. Thank you. Uh, we begin with the uh, adoption of the agenda. Έγκριση μερίσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται. Πάμε στα ανακοινώσεις του Προέδρου, πρώτα απ' όλα τις γλώσσες που έχουμε. Δυστυχώς η διερμηνία έχουμε γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ολλανδικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, σουηδικά, Ογγρικά, λετωνικά, πολωνικά, σλοβακικά, βουλγαρικά, ρουμανικά. Θα τα έχουμε σήμερα, Ευτυχώ μάλλον. Αυτές είναι οι μόνες γλώσσες που έχουμε διερμηνία. Δεύτερον, όσον φάτσε ανακοινώσει του Προέδρου, το Κοινοβούλιο έλαβε σήμερα η θέση του Συμβουλίου στην πρώτη ανάγνωση αφορά την αναθεωρημένο κανονισμό για την Europol σύμφωνα με το άρθρο 66 και παραπέμφθη στην Επιτροπή ταυτόσιμη η θέση του Συμβουλίου του Συμπεφωνημένου κείμενο και επιτρέπει την έγκριση του κειμένου σε πρώιμη φάση τη δεύτερη ανάγνωση. Ο εισηγητή, ο κ. Δία Δεμέρο, προτείνει τα εξή εν ώψη τη δεύτερη ανάγνωση. 20 με 21 Απριλίου συζήτηση του σχεδίου συστάσεω για δεύτερη ανάγνωση στη ΛΥΜΠΕ και καθορισμό προθεσμία για τροπολογίε μόνο στα αγγλικά στι 28 Απριλίου, ψηφοφορία στη ΛΥΜΠΕ, στι συστάσει τη Δευτέρα Αναγνώσεω και στι 10 Νοεμβρίου. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο. 10 Μαΐου ψηφοφορία στην Ολομέλεια στη δεύτερη ανάγνωση. Λοιπόν, πάμε στο σημείο 3 αφορά την έγκριση των πρακτικών. δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θεωρούνται εγκεκριμένα τα πρακτικά. Ωραία. Όλοι έτοιμοι. Προσέχετε. Σημείο 4. Θα ξέρετε από την αλληλογραφία της περισμένης εβδομάδας ότι προσθέσαμε δύο σημαντικά σημεία στη σημερινή μερίσια διάταξη. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο γρήγορος μπορώ. Προσέξτε με λοιπόν. Σημείο 4 και σημείο 5 έξατε σχεδίου συστάσεως για δεύτερη ανάγνωση. Συζητώ με αυτά τα σημεία μετά την απόφαση διάσκεψης των Προέδρων της 7ης Απριλίου να ψηφίσουμε για το πακέτο για την προστασία των δεδομένων και την οδηγία PNR στην Ολομέλεια, την μικρή Ολομέλεια, μήνυ Ολομέλεια Λοιπόν, το Συμβούλιο 8 Απριλίου θέτησε την πρώτη ανάγνωση για το πακέτο τη προστασία των δεδομένων και διαβίβασε το σχετικό κείμενο στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με την νομοθετική διαδικασία που προβλέπεται. Ο πρόεδρο του κοινοβουλίου ανακοίνωσε αρχέ τη ημέρα την έναξη των εργασιών τη Ολομελία, στην αποδοχή όλων των κειμένων παρεπέμφθησαν στην Επιτροπή μα σύμφωνα με το άρθρο 66 που μας επιτρέπει να εξετάσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου για τη δεύτερη ανάγνωση το κείμενο που υπευλήθη από το Συμβούλιο αντιστοιχεί στη συμφωνία που επιταχθεί στις 15 Δεκεμβρίου από Συμβούλιο και Ευρωκοινοβούλιο και Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ενέκρινε τη θέση αυτή στι 17 Δεκεμβρίου. Σα έστειλα επιστολή την περασμένη εβδομάδα και στην επιστολή μου αυτή τη 17η Δεκεμβρίου προ την Προεδρία με την ψηφοφορία Ζήτησα να δούμε αν αντιστοιχεί η θέση του Συμβουλίου στη συμφωνία του κειμένου της 17ης Δεκεμβρίου. Οι νομικοί ε, γλωσσομαθείς, νομικοί, εξέτασαν το κείμενο και δέχθησαν το κείμενο του Συμβουλίου άνευ ε, τοπολογιών για δεύτερη ανάγνωση. Τούτων λεχθέντων, για μια σύντομη παρέμβαση, σύντομες παρεμβάσεις θα δώσω το λόγο στους για τα δύο θέματα και στην Προεδρία του Συμβουλίου για την προστασία των δεδομένων, οδηγία προστασία των δεδομένων. Ε, μπορεί να μας δώσει ε, η κυρία Λόριστον μια παρουσίαση Μάριον. Ευχαριστώ Κλώ, δεν θα επαναλάβω αυτά που ήδη είπες ε, όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου και το ότι είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, διότι έφτασε η μέρα που μπορούμε να έχουμε το πλήρες πακέτο για την προστασία των δεδομένων που θα παρουσιαστεί στην Ολομέλεια και κανονισμό και οδηγία και PNR. Φαντάζομαι ότι αυτές τις μέρες αυτό περιμένει και ο κόσμος από εμά. και χαίρομαι όλους ιδιαίτερος που στη συνεργασία μας αυτή με τους κοιόδης συζητητές όλες οι ομάδες όλοι καταλήξαμε σε αποτέλεσμα το οποίο αποτέλεσμα αυτές τις δύσκολες εποχές θα δείξει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούν μαζί να κάνουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό για να δείξουμε ότι οι ευρωπαϊκές αξίες, θεμελιώδη ανθρωπινά δικαιώματα προστατεύονται, γίνονται σεβαστά και σε πολύ δύσκολες μέρες από τις δυνάμεις της τάξης, την καταπολέμηση της από την τρομοκρατία. Προστατεύουμε και σε αυτή την κατάσταση τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό είναι σημαντικότατο. Και τέλος, εξίσου σημαντικό και στο σημαντικότερο, είδαμε πόσο κρίσιμη είναι η συνεργασία μεταξύ των δυνάμεων της τάξης, Πόσο κρίσιμη η σημασία της ανταλλαγής των πληροφοριών. Και είμαι βέβαιη ότι με αυτή την οδηγία μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα εξελιχθούν πολύ πιο ομαλά τα πράγματα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ Μάριο για την, για το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων. Ο κύριος Άλμπερτ είχε κάποια προβλήματα όσον αφορά τη μεταβασή του. Η Σκά Κέλλερ λοιπόν είχε την καλοσύνη να μας πει μερικά λόγια εκ μέρους του. Λοιπόν, Σκά, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Πράγματι, όπως ανέφερες, τι να κάνει κανείς με την κυκλοφορία και με τα μέσα μεταφοράς. Δεν μπορεί να έρθει ο εισηγητής. Θα έρθει ανα πάσα στιγμή τώρα. Μου ζήτησε όμως να διαβιβάσω το εξή μήνυμα. Και σας λέω αγαπητοί συνάδελφοι, σκιώδεις εισηγητές, μετά από πάνω από τέσσερα χρόνια εργασιών, ε, σαν εισηγητή προτείνω να υιοθετήσετε την πρόταση για τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Όσοι υιοθετήθηκε αυτό και διβιβάστηκε από το Συμβούλιο, είναι αποτέλεσμα εντατικών διαπραγματεύσεων σε φορεί ε, νομοθετικού και στους τριμερείς διαλόγους και στην ψηφοφορία της πρώτης ανάδοσης το Μάρτιο του 2014 και ακολουθήθηκε η γενική προσέγγιση Συμβουλίου από τον Ιούνιο του 2015. Η συμφωνία που εγκατέφθη το Δεκέμβριο επί Λουξεμβριανής Προεδρίας είναι σημαντικό μήνυμα όσον αφορά την ολοκλήρωση του θέματος που, θα που ολοκληρώθηκε από το 2015. Το ανακοίνωσε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και η αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Υιοθετήθηκε την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων τον Δεκέμβριο. Σχεδόν ομόφωνα αυτή η θέση. Αυτό έδειξε ότι βρήκαμε τροστή σωστή ισορροπία. Δηλαδή, θέλαμε υψηλό επίπεδο προστασία για τα θεμελιώδη δικαιώματα στα πλαίσια προστασία των δεδομένων και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών ταυτόχρονα. την άλλη, όμω, θέλαμε να έχουμε μια εύρυθμη ψηφιακή αγορά που θα είναι δίκαιη και να έχει δυνατότητα για καινοτομία και να αναπτυχθεί αυτή η αγορά. Του το να τονίσω ότι δεν πίστευα και δεν πιστεύω ότι αυτές οι δύο πτυχές αποκλείουν η μία την άλλη. Είμαι πεπισμένο ότι σεβασμό τη προσοχή των δεδομένων δεν είναι μόνο προπόθεση για εμπιστοσύνη και για καινοτομία σε μια ψηφιοποιημένη οικονομία, αλλά θα είναι και το κλειδί για την επιτυχία τη οικονομία μα και των οικονομιών μα, μάλλον. Εμεί οι Ευρωπαίοι όχι μόνο εξάγουμε την προστασία τη ιδιωτική ζωή και τα δικαιώματα των καταναλών στο διαδίκτυο, θα κυριαρχούμε στην ψηφιακή αγορά του αύριο, όταν αυτά τα πρότυπα και προδιαγραφέ θα είναι πάρα πολύ σημαντικά για κάθε νέα τεχνολογία, για κάθε προϊόν, για κάθε υπηρεσία. Αυτό ο συμβιβασμό που πετύχαμε μέσω αξιοσημείωτη δημοκρατική διαδικασία τα τελευταία χρόνια, τεράστιο βήμα πρόοδου. Δημιουργούμε μια ενιαία ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την αυριανή ψηφιακή αγορά. Και έτσι εμείς οι Ευρωπαίοι μπορούμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις. Για μία ακόμη φορά, ευχαριστώ τους και ηγητές. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, καθώς και όλους τους εκπροσώπους των διαφόρων συμφερέντων. Ήταν ειλικρινής η προσπάθεια, σκληρή η δουλειά και όλοι συνέβαλαν στο αποτέλεσμα υπό το φως μιας ευρείας συμφωνίας που πετεύθη. Νομίζω ότι η ταχεία διαδικασία εθέτηση του θέματο μαζί με την οδηγία προστασία των δεδομένων αύριο το πρωί σε αυτή την επιτροπή και την Πέμπτη στην Ολομέλεια είναι ο σωστό δρόμο. Όλοι εκεί μα περιμένουν να ολοκληρώσουμε επίσημα τι εργασίε και να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα. Και εκείνοι που ελέγχουν τα δεδομένα, τα κράτη-μέλη και οι σύμβουλοι αυτών έχουν διακαεί πόθο να προχωρήσουν. Το σημαντικότερο, να έχουμε μια ενιαία νομοθεσία την προστασία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή και να υλοποιηθεί. Τη χρειαζόμαστε νομοθεσία. Σήμερα και όχι αύριο. Ευχαριστώ όλους, λέει ο Γιάννη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Οι συγητές στηρίζουν τη διαδικασία λοιπόν που ακολουθούμε. Οπότε παρακαλώ την Προεδρία του Συμβουλίου να πάρει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές και το Συμβούλιο. Χαίρετε πολύ για τη συμφωνία αυτή, που, στην οποία να το Δεκέμβριο που μας πέρασε το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα δύο αυτά θέματα για την προστασία των, της επεξεργασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα. Η συνεργασία μας ήταν πολύ αποτελεσματική και θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του Συμβουλίου, την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και τους συζητητές, την κυρία Λαουριστέν και τον κύριο Άλμπρεχτ, για την επικοδομητική του στάση. Ο κανονισμός για την ε, προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα προστατεύει πράγματι τους ανθρώπους από κάθε κατάχρηση και η οδηγία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας ε, δεδομένων ε, και ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων ακριβώς τον ίδιο στόχο έχει. Αύριο με την ψηφοφορία θα, στη Λίμπε θα μπορέσουμε να ανοίξουμε το δρόμο για να πάει στην Ολομέλεια το θέμα αυτό που είναι και το τελευταίο πολιτικό βήμα προκειμένου οι πολίτες να διαθέτουν τους κανόνες που χρειάζονται σε αυτή τη νέα εποχή για την προστασία των δεδομένων τους. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις σας. Όσον αφορά την διαδικασία, αγαπητοί συνάδελφοι, σα έχω πει σε 7 και 8 Απριλίου, σα ενημέρωσα ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι σήμερα το βράδυ στι 10. Θέλω να σας θυμίσω επίσης ότι μόνο στα αγγλικά θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία, όπως συμφωνήσαν οι συντονιστές της ΛΥΜΠΕ. Οπότε οι τροπολογίες σας πρέπει να κατατεθούν σε μορφή Word και όχι σε e τι 4 τροπολογίες. Και βάσει του άρθρου 66, μόνο τα, οι ευρωβουλευτές ή οι επίσημοι αναπληρωτές μπορούν να υποβάλουν προτάσεις η προθεσμία 11 Απριλίου στι 10 το πρωί για την υποβολή των τροπολογιών. Θα ψηφίσουμε την 3η 12 Απριλίου στι 11 και 4 εδώ σε αυτήν εδώ την ίδια την αίθουσα. Αυτά αγαπητοί συνάδελφοι, αν συμφωνείτε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη τώρα που είναι το θέμα 6. Μια άλλη απώλεια, ένα άλλο θύμα του κυκλοφοριακού. Η συγκεντρική κυρία Βίλστρομ δεν είναι εδώ. Οπότε τι να κάνουμε. Τι λέτε. Θα αργήσει πολύ, ξέρετε. Πέντε λεπτά μου λέτε, μάλιστα. Δεν ξέρω τι να κάνω, λέει ο πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, για να δούμε κυρία Βίλστρομ πότε ακριβώς θα είναι εδώ. Νομίζω ότι καλύτερα να περάσουμε στο επόμενο θέμα, στο πακέτο για την συνοριοφυλακή και εκτοφυλακή. Καλύτερα και να περάσουμε στο θέμα της κυρίας Βίλστρομ μετά. Εντάξει, ωραία. Αγαπητοί συνάδελφοι, λοιπόν, περνάμε ευθύ αμέσω στο σημείο 7 στην ημερήσια διάταξη. Είναι Στρασβούργο, δεν θέλω να σας καθυστερήσω το βράδυ σας πολύ. Εδώ βλέπω φωτογραφίες, selfies, πηγαδάκια. Ωραία, ωραία περνάμε. παρά την ε, χαρά που επικρατεί στην ε, αίθουσα. Σας περάσουμε στο επόμενο σημείο 7. Όλο βλέπω κόσμο να μπαίνει και περιμένω ανυπόμονα να δω την κυρία Βίλστρομ, αλλά όχι. Λοιπόν, σημείο 7, σοβαρό σημείο. Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο φάκελο αυτό για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Εκτοφυλακή αποτελεί προτεραιότητα για μα και μάλιστα είχαμε πολύ λίγο χρόνο να το ετοιμάσουμε το θέμα. Όπω ξέρετε, η φύλαξη των εξωτερικών μα συνόρων είναι προπόθεση για να μην υπάρχουν έλεγχοι στο εσωτερικό των συνόρων μα. Όταν θα έχει εγκριθεί η ρύθμιση αυτή, θα ενισχυθούν τα εξωτερικά μα σύνορα και θα αντιμετωπιστούν διάφορε αδυναμίε που έχουν εντοπιστεί τώρα όσον αφορά τη ρύθμιση της Frontex. Ο κύριος Πάπριξ θα μας παρουσιάσει το σχέδιο πρότασής του. Είναι έτοιμος? Ναι, από ό,τι βλέπω. Μετά τον εισηγητή θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Προεδρία 10 λεπτό καθένας το πολύ. Και μετά θα ζητήσω από τον κύριο Λεγκέρη και τον κύριο Βιβυρόφσκι για περίπου 7 λεπτό καθένας να πάρουν το λόγο. Και στη συνέχεια θα συζητήσουμε το θέμα με τους σκιώδες εισηγητές και με όποιον άλλον Ευρωβουλευτή το επιθυμεί. Οπότε, περνάμε στον κύριο Πάμπριξ. Παρακαλώ κύριε Πάμπριξ να μας παρουσιάσετε το σχέδιο έκθεσή σας και συγγνώμη που αλλάξαμε τη σειρά των θεμάτων. Είσαστε έτοιμος κύριε Πάμπριξ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, για μένα είναι μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που μπορώ να σας παρουσιάσω την έκθεσή μου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Εκτοφυλακή. Όπως είπατε και εσείς ε, νωρίτερα, την πρόταση αυτή την πήραμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από λίγο σχετικά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και εγώ και οι σκιαώδεις εισηγητές αναγκαστήκαμε να περιοριστούμε λόγω χρόνου. Θέλω να πω δύο λόγια όμως και για την μορφή χαίρομαι πραγματικά που μπορέσαμε να δουλέψουμε με διαφάνεια με τους εκπροσώπους των άλλων πολιτικών ομάδων εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τους σκιώδεις εισηγητής από όλες τις ομάδες. Η συνεργασία ήταν πολύ επικοδομητική. Αποτέλεσμα είναι το σχέδιο αυτό έκθεσης που σας το παρουσιάζω σήμερα. Λοιπόν, είναι περιδό νομίζω να υπογραμμίσουμε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικός είναι ο χώρος Σέγγεν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο σημαντικός είναι για όλους μας και πόσο σημαντικό είναι για όλους μας να αντιμετωπίσουμε την μεταναστευτική και προσφυγική κρίση σήμερα στην Ευρώπη. Όσον αφορά το Σέγγεν, είναι ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα, ακριβώς επειδή τα εξωτερικά μας σύνορα βρίσκονται υποπίεση, κινδυνεύουμε όλο και περισσότερο να απαρατηθούμε από κάτι τόσο σημαντικό όπως είναι ο χώρος έγκεν. Για να μην συμβεί λοιπόν αυτό, είναι σημαντικό να προχωρήσουμε με βελτιώσεις όσον αφορά τη διαχείριση των εξωτερικών μας συνόρων και τη φύλαξή τους. Και φυσικά ο χρόνος εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων αποτελεί προϋπόθεση όχι μόνο για να βρούμε καλύτερες λύσεις στη μεταναστευτική κρίση από την οποία όλοι υποφέρουμε σήμερα, αλλά και για να διασφαλίσουμε μεγαλύτερη προστασία των χωρών μας και των πολιτών μας. Όλοι ξέρουμε για τις τραγικές επιθέσεις, τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες, αλλά θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Μεταξύ άλλων και γι' αυτό λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κάτι για να διασφαλίσουμε την προστασία μας. Όσον αφορά τώρα κάποιες αρχές που περιλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο έκθεσης. Πρέπει να αναφέρω πρώτα απ' όλα ότι έχουν ακουστεί διάφορες επικρίσεις από αυτούς οι οποίοι φοβούνται ότι εφόσον υπάρξει περισσότερη συνεργασία όσον αφορά τη διαχείριση της φύλαξη των συνόρων, αυτό θα οδηγήσει σε μείωση της κυριαρχία των χωρών μελών. Δεν είναι αλήθεια όμως αυτό, γιατί αν δείτε το σχέδιο το οποίο ετοιμάσαμε συλλογικά και σας το υποβάλλουμε σήμερα προς παρετέρω βελτίωση, η συνοριοφυλακή και εκτοφυλακή αυτή ευρωπαϊκή ενισχύει την κυριαρχία των χωρών μελών διότι η Ευρώπη είναι τόσο δυνατή όσο δυνατά είναι τα επιμέρους μέλη της. Οπότε φυσικά και χρειάζεται σύρρηξη σε όλες τις χώρες και αυτό σημαίνει ότι ενισχύεται η ίδια ικανότητα των χωρών μελών από την κοινή αυτή προσπάθεια. Επίσης θέλουμε να διασφαλίσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες για το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα αποτελεσματικό σχέδιο. Ίσως δεν τα έχουμε καταφέρει με όλες μας τις πολιτικές αποφάσεις μέχρι τώρα. Κάθε φορά δεν μπορώ να πω ότι είμαστε πάντα περήφανοι για την αποτελεσματικότητά μας. Τώρα όμως αυτή η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Εκτοφυλακή αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα για βελτίωση, βελτίωση της Frontex και βελτίωση της αποτελεσματικότητά μας. Ώστε είμαστε καλύτεροι δηλαδή από ό,τι είμαστε κατά το παρελθόν στη διαχείριση των εξωτερικών μας συνόρων. Οι πολίτες μας λοιπόν χρειάζονται περισσότερη ασφάλεια οι πολίτες μας πρέπει να πιστέψουν ε, και να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε βασισμένοι σε δύο αρχές. Η μία αρχή είναι εκείνη που λέει ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να αγκιάται ότι ο οργανισμός αυτός θα είναι πιο αποτελεσματικός από ό,τι είναι σήμερα η Frontex. Η δεύτερη πρόκληση που είχαμε όλοι μπροστά μας ήταν ε, ο χρόνος που πίεζε. Διότι αν πιεστούμε υπερβολικά όσον αφορά το χρόνο, τότε κινδυνεύουμε να μην πάρουμε και τις σωστές αποφάσεις για να αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό, το προσφυγικό κλπ. Δεν μπορούμε να περιμένουμε περισσότερο, γιατί δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε κανένα άλλο επίπεδο αν δεν έχουμε φροντίσει για την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων. Προσπαθήσαμε λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας, βάσει των δύο αυτών αρχών, όλες τις προτάσεις που μας ερχόντουσαν από τις διάφορες πολιτικές ομάδες και τους σκιώδες εισηγητές, οι οποίοι συμφώνησαν στη βασική ιδέα τελικά της πρότασής μας. Τα πιο επίμαχα ζητήματα στην έκθεση αυτή ποια είναι. Το ένα είναι η εθνική κυριαρχία. Σας το είπα ήδη. Το δεύτερο είναι Τι κάνουμε αν μια χώρα μέλη δεν θέλει να συνεργαστεί, ακόμα και αν πιέζεται από μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Εδώ νομίζω ότι καταφέραμε να βρούμε ένα καλό συμβιβασμό για το πώς μπορούμε χωρίς να πλήξουμε την εθνική κυριαρχία των χωρών μελών, να βρούμε τρόπο ώστε να μην πληγεί η ευρωπαϊκή κυριαρχία. Υπάρχει μια πολύ καλή πρόταση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει να υπάρξει μια εφεδρεία με 1.500 συνοριοφύλακες, αλλά εκεί να υπάρχουν επιπλέον και κάποιοι πυρογνώμονες, οι οποίοι να σταλούν στη χώρα που βρίσκεται σε κρίση. Και μάλιστα δεν θα το έλεγα ε, εφεδρεία, θα έλεγα ταχείας αντίδρασης. Αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να είναι έτοιμοι να βρεθούν εκεί που υπάρχει κρίση. Και σε αυτήν την δύναμη τη ταχείας αντίδραση θα συμμετέχουν όλε οι χώρε που έχουν εξωτερικά σύνορα. Ένα άλλο θέμα είναι οι αξιωματούχοι, σύνδεσμοι αξιωματούχοι, οι αξιωματικοί σύνδεσμοι. Και αυτούς πρέπει να τους λάβουμε υπόψη μας, να μην υπάρχουν διακρίσεις. Και βέβαια αυτό που έχει τεράστια σημασία είναι η τάχιστη ανταλλαγή πληροφοριών. Ο οργανισμός αυτός μπορεί να βοηθήσει λοιπόν τις χώρες μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα και αυτό με διάφορα εργαλεία. Γιατί θα έχει και τεχνική αρρωγή να προσφέρει. Αν κάποια χώρα αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ή βρίσκεται σε αδύναμη κατάσταση, οι τεχνικοί υπερογνώμονες μπορούν να βοηθήσουν να προσφέρουν αυτή την τεχνική αρρωγή και στον τομέα της έρευνας και στον τομέα της διάσωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως πρέπει να δείξει ότι είναι αποτελεσματική. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι πολύ βασικό αυτό. Πάνω στην αποτελεσματικότητα έχει χτιστεί ολόκληρο το οικοδόμημα. Ο οργανισμός αυτός επίσης διαθέτει και διάφορες ρήτες ασφάλειας όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα του, για την προστασία του κάθε ανθρώπου που μπορεί να εμπλακεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο έργο του οργανισμού αυτού. Απαιτείται λογοδοσία από τον οργανισμό και εδώ συμμετέχουν και το Συμβούλιο και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Και το Κοινοβούλιο έχει και αυτό να παίξει ρόλο στην επιλογή του επικεφαλής του οργανισμού, για παράδειγμα, του εκτελεστικού διευθυντή και γενικά των ε, ανθρώπων που θα είναι επικεφαλής στον οργανισμό αυτό. Αν λοιπόν καταφέρουμε να πετύχουμε, να δημιουργήσουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Συνοριακή ε, και Ακτοφυλακή, έγκαιρα, αυτό θα είναι μεγάλη επιτυχία για μας. Θα ανακτηθεί η ελπίδα, αλλά και η πίστη πολλών Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι η προστιθέμενη αξία που έχει αναλάβει στους ώμους της αυτή η νέα υπηρεσία, αυτός ο νέος οργανισμός. Θέλω επίσης να υπενθυμίσω ότι δεν πρέπει να νομίζουμε ότι ο οργανισμός αυτός θα μας λύσει όλα τα προβλήματα χρειάζεται χρόνος και αποφάσεις σε πολλές άλλες υποθέσεις. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν το έγγραφο αυτό με όλες τις με όσα αναφέρει, να μην το φορτώσουμε με κάθε ιδέα που περνάει από το κεφάλι μας. Έχουμε χρονοδιάγραμμα, έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις που προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε όσο γίνεται περισσότερο και όχι με καλές προθέσεις να καταστρέψουμε ένα καλό έργο που έχει ήδη γίνει. Μέχρι τώρα έχουμε δουλέψει με όλους τους σκιώδεις και τους εμπειρογνώμονες από τα άλλα θεσμικά όργανα και πιστεύω ότι έτσι μπορούμε να πετύχουμε. Ελπίζω τους επόμενους μήνες να έχουμε την απόδειξη και από τις άλλες πολιτικές ομάδες ότι θα στηρίξουν το έγγραφο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ας πάμε κατευθείαν στην Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσω με αυτά που συμπέρανε και ο εισηγητής ότι αυτή η πρόταση για τη συνοριοφυλική και την αγροφυλακή δεν είναι πανά και δεν θα ε, επιλύσει όλα τα προβλήματα που συνδέονται με την μεταναστευτική κρίση υπάρχει ένα σύνολο μέτρων που έχουν ε, προταθεί, κάποια έχουν εγκριθεί, κάποια έχουν εφαρμοστεί, κάποια όχι. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σύνολο μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να έχουμε μία σωστή ανταπόκριση στην μεταναστευτική κρίση με όλες τις πτυχές της. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον εισηγητή και επίσης και το Συμβούλιο που αντέδρασαν τάχιστα σε αυτό το θέμα, ώστε σήμερα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να έχουμε το σχέδιο του κυρίου Πάμπριξ, κάτι απαραίτητο, γιατί για να διασφαλίσουμε το Σέγγεν θα πρέπει να επανακτήσουμε τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Και να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι κάνοντας λόγο για την επανάκτηση του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε μόνο να κρατήσουμε τους πρόσφυγες απ' έξω, αλλά να αποφασίσουμε αν κάποιος δικαιούται να εισέλθει και για αυτούς που δεν έχουν αυτό το δικαίωμα να τους κρατήσουμε εκτός των συνόρων. Άρα δεν δημιουργούμε ένα φρούριο Ευρώπη, μια Ευρώπη φρούριο, απλώς θα βελτιώσουμε τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων ως μέρος ενός πιο αποτελεσματικού ελέγχου της μετανάστευσης. Να ευχαριστώ τον κύριο Πάμπριξ και τους ε, σκιώδες ηγητέ για τις επικοδομητικές συναντήσεις που είχαμε μέχρι τώρα. Και από ό,τι φαίνεται είναι όλοι πρόθυμοι να εργαστούν ε, με ταχύτητα σε αυτό το ουσιαστικό ζήτημα. Γνωρίζω ότι και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο υπάρχει ευελιξία και αυτό είναι σαφές και στην έκθεση του κύριου Πάμπριξ. Θεωρώ ότι οι δύο συνομοθέτες είναι έτοιμοι να ρεχθούν σε ένα πνεύμα ε, συνεργασίας. Είναι κάτι που χρειαζόμαστε πηγόντως για να αποτέψουμε και στο μέλλον ε, παρόμοιε μεταναστευτικέ κρίσει που ενδεχομένω θα αντιμετωπίσουμε. Μία πτυχή στην οποία θέλω να πιστήσω το ενδιαφέρον σα είναι ότι πρόσφατα λάβαμε την γνωμοδότηση του ε, Ευρωπαίου Πόπτη για την Προστασία των Δεδομένων, γιατί η ταχύτητα με την οποία εργάζεται η Επιτροπή και παρουσιάζει αυτή την πρόταση Χρειαζόμασταν μια εκ των προτέρων διαβούλευση με τον επόπτη. Από ό,τι βλέπω όμω και ο εισηγητής και η Προεδρία στο κοινό κείμενο που εξεδόσαν έχουν λάβει υπόψη τις συστάσεις που έχουν γίνει από τον Ευρωπαίο Πόπτη Προστασίας Δεδομένων και έτσι και οι τρεις από κοινού μας δείχνουν ε, και μάλλον δύο και Συμβουλίο πρέπει Επιτροπή δείχνουν πώ μπορούμε να λάβουμε υπόψη ε, τι τάσει του επόπτη προστασία δεδομένων. Άρα δεν αποτελεί έκπληξη ότι και στην έκθεση του κ. Βαμπρίξ αλλά και στον έγραφο του Συμβουλίου τα ίδια θέματα ε, θίγονται όπως είναι η αξιολόγηση τροτότητας, η αξιολόγηση του μηχανισμού Σέγγεν, η υποχρεωτική συνεισφορά των κρατών μελών και για την παροχή πόρων και τεχνικού εξοπλισμού στην, στον οργανισμό ώστε να μπορέσει να αναλάβει δράση ο οργανισμός. Για να μιλήσω λίγο πιο απλοϊκά, στο Συμβούλιο για τη διάρκεια των συζητήσεων υπήρχε μία τάση ε, για την παρουσία περισσότερων κρατών μελών στην ε, ε, δημιουργία της νεοφιλικής και της εκτοφυλακής. Στην έκθεση που παρουσιάστηκε σήμερα από τον κύριο Πάμπριξ, υπάρχει περισσότερη παρουσία του Κοινοβουλίου, η λογοδοσμότητα του οργανισμού, ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην ε, ε, στο διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και για να σας δώσω ένα παράδειγμα στην αξιολόγηση τροτότητας ε, στο συμβαστικό έγγραφο του Συμβουλίου αναφέρεται ότι θα πρέπει να, πρέπει να υπάρχει αυτή η αξιολόγηση τροτότητας και να σχολιαστεί και επίσης στην έκθεση του κ. Πάπληξη είναι και πάλι αναφορά ε, σε αυτή την αξιολόγηση τροτότητας. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια συμβατότητα. Όταν θα έχουμε μια ολοκληρωμένη θέση από την πλευρά της ΛΥΜΠΕ, θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε και μια ισορροπία ανάμεσα στους, στα όργανα, στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο. Όμως από ό,τι φαίνεται είναι δυνατό να φτάσουμε σε μια συμφωνία που θα είναι ικανοποιητική για όλους. Θα ήθελα επίσης να σας πληροφορήσω ότι στο Συμβούλιο έχουμε συμμετάσχει στο διάλογο, επικοδομητικά όπως και εδώ. Έχουμε μια κοινή προσέγγιση προς αυτό από την πλευρά του Συμβουλίου και να σας ε, πω ότι η Επιτροπή αποδέχθηκε και να έκρινε όλες τις ε, τροπολογίες που προτάθηκαν από το Συμβούλιο. Φυσικά θέλουμε να ακούσουμε για την θέση του Κοινοβουλίου και στη συνέχεια θα ε, οριστικοποιήσουμε και εμείς τη θέση μας με ενδεχόμενες αλλαγές της ε, πρότασης. Έτσι λοιπόν ανυπομονούμε να ακούσουμε και τους γεώδεις εισηγητές, τις δικές τους ε, απόψεις για το σχέδιο του κύριου Πάμπριξ και είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε στον τρίλογο ώστε να βρούμε το στομότερο δυνατό μια λύση. Ευχαριστώ. Ο, ο κύριος Λούστερμπεργκ, εκπρόσωπος της Προεδρίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στο Στρασβούργο να είμαστε παρόντες στην παρουσίαση σχεδίου έκθεσης. Να ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Πάμπρεξ και τους ε, σχιώδεις εισηγητές για τη συνεργασία που είχαμε σε αυτό το φάκελο. Φυσικά να μην ξεχάσω και την Επιτροπή, τη οποία συνεργασία ήταν επίσης πολύτιμη. Για το Συμβούλιο δεν αποτελεί εκπλήξη ότι αυτό ο φάκελο θεωρείται προτεραιότητα. Εξαιτία τη κατάσταση στα εξωτερικά σύνορα υπήρξε μια σαφή προθεσμία από την Προεδρία ε, το Φεβρουάριο και αποφασίστηκε ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε τις εργασίες σε αυτό το φάκελο για να καταλήξουμε σε μια απόφαση στο τέλος του εξαμήνου. Και αυτό δείχνει τη δέσμευσή μας ως προς ε, την επίτευξη συμφωνίας. Χαίρομαι για το γεγονός ότι και τα άλλα θεσμικά όργανα έχουν την ίδια δέσμευση. Στο Συμβούλιο επιταχύναμε τις εργασίες μας και αυτό έχει ως αποτελέσμα να επιτευχθούν συμφωνίες στο κείμενο σε επίπεδο την προηγούμενη εβδομάδα. Με αυτές τις συμφωνίες η Προεδρία έχει την εντολή από το Συμβούλιο να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο και ανυπομονούμε ε, να ξεκινήσουμε φυσικά. Όπως ε, η Επιτροπή και ο Συγητής, σε σχέση με το περιεχόμενο θα πω και εγώ ότι υπήρξαν πολύ σημαντικά θέματα για το Συμβούλιο αλλά και η πρόταση τη Επιτροπή ήταν μια πάρα πολύ καλή ε, βάση. Καταφέραμε να κρατήσουμε τα βασικά στοιχεία της πρόταση τη Επιτροπής ε, στο έγγραφο, στο κείμενο του Συμβουλίου. Οι πιο σημαντικέ αλλαγέ είχαν να κάνουν με την ε, κοινή ευθύνη και την αξιολόγηση των τρότητας όπου θεωρήθηκε ότι η διαχείριση των εξωτερικών ε, συνόρων είναι η κοινή ευθύνη των κρατών μελών και πράγματι στη δικασία οδηγηθήκαμε στην αξιολόγηση τροτότητας για να υπάρξουν παρεμβάσεις και να και παίξει σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων και το Συμβούλιο. Αναφέρθηκε ένα ακόμα στοιχείο από τον εισηγητή, αν κάποιο δεν θέλει να ακολουθήσει ε, την απόφαση αυτή που έχει ληφθεί και σε αυτό το θέμα βρήκαμε μία λύση σε σχέση με την ε, εθνική κυριαρχία των κρατών μελών, μία λύση που είναι επίσης πολύ αποτελεσματική. Όσον αφορά τα υπόλοιπα σημαντικά θέματα, η προστασία των δεδομένων, οι ρήτρε ε, που έχουν τεθεί στην πρόταση της Επιτροπής καταφέραμε να τα λάβουμε υπόψη να λάβουμε υπόψη ανησυχίε που αφορούν ε, την προστασία των δεδομένων ε, προσωπικής, προσωπικού χαρακτήρα. Είναι ένα θέμα αυτό στο οποίο καταλήξαμε στη συμφωνία στα τέλη Μαρτίου. Επίσης, ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μα με τον εισηγητή και του κοιόδης εισηγητή και με την Επιτροπή με στόχο την επίτευξη συμφωνίας σε αυτό το φάκελο. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Λετζέρη από τη Frontex έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να αναφερθώ σε επιχειρησιακές μου εμπειρίες. Καταρχάς, θέλω να αναφερθώ στην εντολή που εμπεριέχεται στην πρόταση. Μετά θέλω να αναφερθώ στη λογοδοσία, στον έλεγχο. Όλο βασίζονται στην εμπειρία του οργανισμού. Οι επιχειρησιακές προπτικές και σαν εκτελεστικός διευθυντής τα τελευταία, τελευταίους 15 μήνες ε, είδα κάποια πράγματα και συνελέξα εμπειρίες. Όσον αφορά την εντολή, όπως και άλλοι ομιλητές, επιβεβαίωνω ότι είναι σημαντική αξιολόγηση βαλωτότητας των κρατών μελών και είναι σημαντικό να είναι αυτόνομος οργανισμός στην εκτέλεση του έργου του. Γι' αυτό κάνουμε αξιολόγηση του κινδύνου τώρα. Θα πρέπει ο φορέας να έχει τη δυνατότητα να κάνει την αξιολόγηση του πόσο ευάλωτη είναι μια χώρα. Όσον αφορά τις δυνατότητες που έχουμε, είδαμε πέρσι να. Ήταν σαφές ότι τα κράτη-μέλη, ο οργανισμός και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόταν περισσότερες δυνατότητες, περισσότερους μεθοριοφύλακες, περισσότερο εξοπλισμό. Όλα αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν χωρίς χρονοτριβή στα εξωτερικά σύνορα. Είναι σημαντικότατο να υπάρχει δυνατότητα να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει προσωπικό να μπορεί να αντιδράσει σε περίπτωση ανάγκης. Και ο φορέας να έχει τον εξοπλισμό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το κείμενο που έχουμε μπροστά μας. Θα σας δώσω και ένα παράδειγμα. Να σας πω τι έγινε το τελευταίο μήνα από πλευράς Frontex. Αποκτήσαμε τη δυνατότητα να μισθώνουμε αεροσκάφη ή και να αγοράζουμε υπηρεσίες εναερίου ελέγχου. Χρησιμότατο αυτό. Έτσι μπορούσαμε να ξεπεράσουμε κάποια προβλήματα όταν δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν τα κράτη-μέλη, όταν δεν είχαν ε, αέρια μέσα για τον έλεγχο. Επίσης είναι σημαντικό να υπάρχει στατικικός συντονισμός μεταξύ κρατών μελών. Ο οργανισμός θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο. Παραδείγματος χάρη, η Frontex δεν ενημερώνεται για τα σχέδια των κρατών μελών, δηλαδή δεν ξέρει αν τα κράτη-μέλη θέλουν να κάνουν περικοπές στον φάρτο προσωπικό όσον αφορά τον αριθμό των μεθοριοφυλάκων. Δεν γνωρίζει ο φορέας μας και πώς αναπτύσσονται οι μεθοριοφύλακες σε κάθε χώρα. Ποια είναι τα σχέδια της κάθε χώρας. Άρα η Frontex αυτό μπορεί να το βελτιώσει. Να βελτιώσει το συντονισμό των χωρών. Πράγματι, ο οργανισμός δεν ασχολείται μόνο με τα μεταναστευτικά θέματα, αλλά όπως είδαμε και πέρσι από τα γεγονότα, υπήρχε και ε, δεν έπρεπε να έχουμε απομονωμένα δοχεία στον αφάς πληροφορίες. Ούτε διαχωρισμοί μεταξύ πρώτου και τρίτου πυλώνα πρέπει να υπάρχουν. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Νοεμβρίου, το Συμβούλιο Εσωτερικών και Δικαιοσύνης ζήτησε από τους διάφορους φορείς και από τη Frontex να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη όσον αφορά τα κέντρα υποδοχής, τα hotspots. Να ένα παράδειγμα. Εντός τη φυστάμενη εντολής αναπτύξαμε καλύτερη συνεργασία με την Ευρωπόλ και με τις δυνάμεις της τάξης. Και εδώ έρχομαι στα προσωπικά στοιχεία. Ευαίσθητο θέμα. Έχουμε φιλόδοξη πρόταση. Να πω απλώς το εξής. Ο οργανισμός στηρίζει τα κράτη-μέλη όσον αφορά τα hot spots. Και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Μεθοριοφυλοκής που αναπτύσσονται στα κράτη-μέλη για να είναι αποτελεσματικοί στο έργο τους θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν και βάση δεδομένων όπως είναι το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν το σύστημα πληροφοριών θεωρήσει και βάσεις δεδομένων που βοηθούν εκείνους που ελέγχουν τα σύνορα. Και αυτό πρέπει να γίνει στο μέλλον. Έτσι όλα θα είναι πιο διαφανή και πιο εύκολα. Αν ο οργανισμός μας μπορεί να έχει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων. Βέβαια, έλεγχος πρέπει να υπάρχει, πλήρης παρακολούθηση, του τρόπου χρήσεως των προσωπικών δεδομένων. Να πω και κάτι άλλο. Συνεργασία με άλλους φορείς εσωτερικών και δικαιοσύνης. Αναφέρθηκα στη συνεργασία με την Ευρωπόλ. Βελτιώθηκε αυτή. Π.χ. μέσω των διαφόρων σχεδίων που εφαρμόζονται στα πλαίσια της επιχειρήσεως τρίτων στην Ιταλία και θα επεκταθεί αυτή η συνεργασία. Να πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Frontex και που διαβιβάζονται σε, άλλες, σε άλλους φορείς των οργάνων της τάξης. Πρέπει να συνεργαστούμε και με την ΕΑΖΟ. Χρειάζεται ισορροπημένη διαχείριση των συνόρων. Η Frontex είναι έτοιμη να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και αν βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο, τότε και εμείς θα μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα με τους άλλους φορείς. Η ακτοφυλακή τώρα. Φέτος ο οργανισμός μας θα δώσει πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ για θαλάσσιες επιχειρήσεις. Είναι και το μεγαλύτερο βήμα πρόοδο αυτό αν τελικά καταφέρει ο οργανισμός μας να αναπτύξει τη συνεργασία με την ακτοφυλακή επισήμως και με άλλους φορείς της τάξεως και τα τελωνία. Συνεργαζόμαστε με τους άλλους φορείς όπως την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου Τσαλίας ή την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια των Θαλασσίων Μεταφορών. Εφαρμόζουμε πιλωτικά προγράμματα. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι στο μέλλον θα είναι Σημαντικότατε οι προσπάθειε στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Δηλαδή, η Frontex να μπορεί να συνεργάζεται καλύτερα με τι ακτοφυλακές και με τους διάφορου φορεί για την ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών. Κάποια σχόλια έχω τώρα όσον αφορά τον έλεγχο και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Βασίζομαι στην προσωπική μου εμπειρία σαν εκτελεστικός διευθυντής της Frontex, σε αυτά που σας λέω. Είναι κρίσιμο ένας οργανισμός όπως η Frontex να γίνεται αντιληπτή ως φορέας ε, υποδημοκρατικό έλεγχο που λογοδοτεί. Γι' αυτό προσεκλήθη επανειλημμένο σε αυτή την Επιτροπή. Αλλά και σε άλλες Επιτροπές στο Κοινοβούλιο. Καμιά φορά προσεκλήθην και από εθνικά κοινοβούλια. Και οπότε ήταν δυνατόν να γίνει αυτό, ήταν πολύ επικοδομητικό να απαντήσει ο οργανισμός μας ερωτήσεις και να ελέγχεται. ελεγχόμεθα και από τον Εποπτικό Φορέα την προστασία των δεδομένων, τον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Μας βοηθάει αυτό, διότι ο οργανισμός μας μπορεί να συμμορφώνεται έτσι με τις συνθήκες, με το πλαίσιο του νόμου, με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Επιβεβαιώνω ως εκτελεστικός διευθυντής ότι αισθάνθηκα την ανάγκη να αποδείξω ότι ο οργανισμός μας είναι διαφανής, <clears throat> διαφανής και ελεγχόμενος. Κλείνοντας, είναι κοινή ευθύνη, είναι ευθύνη κρατών μελών και του οργανισμού μας. Καμιά φορά είναι δύσκολο τα κράτη-μέλη και τα άλλα θεσμικά όργανα το κατανοήσουν αυτό. Είναι όμως τομέας δραστηριοτήτων βλέπετε που ως εκτελεστικός διευθυντής αναμένω σαφήνεια. Έτσι είμαι σίγουρος ποιος είναι υπεύθυνο για συγκεκριμένα πράγματα. Ποιος λογοδοτεί σε ποιον. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, των κοινών επιχειρήσεων, η ευθύνη, η λογοδοσία πρέπει να είναι ξεκάθαρα πράγματα. Είναι σημαντικό θέμα αυτό. Έτσι μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Κύριε Λιτζέρη, σας παρακαλώ παραμείνετε να ακούσετε και τους σκιώδεις εισηγητές και τους ευρωβουλευτές τι έχουν να πούνε, γιατί ο ρόλος της ΦΝΟΤΕΚ σίγουρα είναι πολύ σημαντικός και καλό θα ήταν να μείνετε για να ακούσετε τη συζήτηση. Τώρα, πριν να δώσω το λόγο στους επόμενους, ας ακούσουμε τον κύριο Βιρεγδρόσκι, ο οποίος είναι εκ μέρους του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω και να παρουσιάσω στην Επιτροπή σας τα κύρια συμπεράσματα και κάποιες συστάσεις του επόπτη προσωπικών δεδομένων που είναι η αρχή, η αρμόδια για αυτά τα θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η άποψη του Ευρωπαίου επόπτη έχει υποβληθεί ήδη από το Μάρτιο έτσι όπως ε, προτάθηκε από την Επιτροπή του Δεκέμβρη που μας πέρασε. Ο κύριος Μπουταρέλη λοιπόν, ο επόπτης Ευρωπαίος Προσωπικών Δεδομένων και εγώ ο ίδιος, κοιτάξαμε τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να μπορεί να πετύχει η πρωτοβουλία αυτή για την συνοριοφυλακή και την ακτοφυλακή. Εξετάσαμε νομικά λοιπόν το θέμα και Είπαμε ότι πρέπει να στηρίξει και το κοινό τις δραστηριότητες αυτές του νέου οργανισμού. Η προσφυγική κρίση και οι τρομοκρατικές επιθέσεις ε, πέρυσι στη Γαλλία και πριν από λίγο στις Βρυξέλλες οδήγησαν τη, στο να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα περισσότερο σε πίεση και να πρέπει να υιοθετήσει μέτρα για να διαχειριστεί καλύτερα τον έλεγχο των συνόρων της και να προστατεύσει καλύτερα τους πολίτες της για να μην νιώθουν το φόβο που έχει μπει στις ζωές τους. Η καταπολέμηση τρομοκρατίας, εγκλημάτων, αντιμετώπιση του προσφυγικού είναι τα κύρια, ε, κύριοι στόχοι σχετικά με τους οποίους πρέπει να αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, ο επόπτης ε, Ευρωπαίος Δεδομένων δεν είναι ο πρώτος ο οποίος θα μιλήσει για τα μέτρα εκείνα τα οποία ε, πρέπει να ληφθούν. Όμως, ο ρόλος της αρχής αυτής είναι να αναγκάσει εκείνους που παίρνουν αποφάσεις να εξηγήσουν γιατί παίρνουν τέτοια μέτρα ελέγχου των πολιτών, για παράδειγμα, και να τους καταδείξουμε πως μερικές φορές τα μέτρα αυτά μπορεί να είναι δυσανάλογα με το στόχο. Ο κανονισμός τώρα, τον οποίο συζητάμε σήμερα, μπορεί πράγματι να παρέμβει στα... και να παραβιάσει τα δικαιώματα κυρίως προσφύγων και μεταναστών που είναι και πιο ευάλωτες ομάδες ανθρώπων που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας. Από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γνωρίζουμε ήδη και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εφαρμόζει τις αρχές της Χάρτας Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε περιπτώσεις όπως αυτές και ξέρουμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Η γνωμοδότησή μας αναφέρει πέντε ανησυχίες του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και κάνει κάποιες συστάσεις προκειμένου ο κανονισμός αυτός να συμμορφωθεί απόλυτα με τις αρχές του Ευρωπαίου Επόπτη. Ήδη είχαμε διάφορες συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ολλανδική Προεδρία προκειμένου να συζητήσουμε την πρόταση και να βρούμε τρόπους να ενσωματώσουμε τις συστάσεις αυτές στο κείμενο. Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ και πέρυσι την Frontex ε, δύο φορές και συναντήθηκα με τον κύριο Λετζέρη και στις Βρυξέλλες. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, οι ανησυχίες μας έχουν να κάνουν με το διτό στόχο της πρωτοβουλίας αυτής, δηλαδή διαχείριση μετανάστευσης αφενός και ασφάλεια και επιβολή του νόμου αφετέρου. Πρέπει να υπάρχει σαφής ορισμός των στόχων αυτών, προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά το κατά πόσο τηρούνται οι αρχές προστασίας δεδομένων όπως πρέπει. Πρόκειται για δύο στόχους που απαιτούν διαφορετική αξιολόγηση για την αναγκαιότητα, την αναλλαγικότητα κλπ. Συστήνουμε λοιπόν περισσότερες λεπτομέρειες και χωριστή αντιμετώπιση των δύο αυτών στόχων για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της δράσης. Η αναλογικότητα, για παράδειγμα, πρέπει να μετριέται εκ των προτέρων να ξέρουμε γιατί συλλέγονται τα δεδομένα και γιατί χρησιμοποιούνται. Με τι σκοπό. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι εφικτό να υπάρξει καλή ισορροπία ανάμεσα στον έλεγχο της αυξηνόμενης μετανάστευσης, της ανάγκης για περισσότερη ασφάλεια, αλλά και την προστασία των μεταναστών και των προσφύγων. Όμως προς το παρόν δεν γνωρίζουμε να έχει υπάρξει ιδιαίτερη πρόοδος επ' αυτού στον προτινόμενο κανονισμό. Οπότε επαναλαμβάνουμε τη σύστασή μας αυτή. Τώρα, για να υπάρχει νομική βεβαιότητα και διαφάνεια, συστήνουμε διευκρίνηση του εύρους των δραστηριοτήτων συλλογής ε, δεδομένων και άλλων λειτουργιών του νέου οργανισμού. Θα έπρεπε να υπάρχουν κατάλογοι που να αναφέρουν εκτενώς τις διάφορες κατηγορίες δεδομένων που θα χρησιμοποιούνται και που θα περνάνε από άλλες αρχές στον οργανισμό αυτό. Επίσης πρέπει να είναι σαφής ποιες είναι οι αρμοδιότητες του νέου οργανισμού, τον οποίο θα εποπτεύει ο Ευρωπαίος Επόπτης Προσωπικών Δεδομένων και από την άλλη μεριά ποιος θα είναι ο έλεγχος των χωρών μελών. Δηλαδή να ξέρουμε πώς ακριβώς λογοδοτεί ο νέος αυτός οργανισμός. Χαίρομαι πάντως που και ο συγγετής ο κύριος Πάμπριξ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρουν το θέμα της λογοδοσίας και ο κύριος Λεγκέρη επίσης το ανέφερε στην παρουσίασή του. Οι προποθέσει κάτω από τις οποίες συλλέγονται τα δεδομένα στα σύνορα από τις χώρες μέλη και που θα πηγαίνουν μετά στον οργανισμό σημαίνει ότι ο έλεγχος πρέπει να ορίζεται καλύτερα και το ποιος κάνει τον έλεγχο αυτό. Και χαίρομαι που ο κύριος Λετζέρη ζήτησε το ίδιο. Για την μεταβίβαση τώρα τέτοιων προσωπικών δεδομένων εκτό Ευρωπαϊκή Ένωσης και εδώ έρχομαι στην τέταρτη ανησυχία μας. Πρέπει να δούμε πώς θα γίνεται η μεταβίβαση αυτή εφόσον πρόκειται για επιστροφή των μεταναστών ή προσφύγων στην χώρα προέλευσής τους. Και τέλος, ρήτρε προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στην πρόταση. Εδώ θέλω να πω ότι τα άτομα των οποίων τα δεδομένα ε, μεταβιβάζονται πρέπει να ενημερώνονται, όπως επίσης πρέπει να ενημερώνονται και τα δικαιώματά τους. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να δίνονται από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες τόπου, με τον σωστό τρόπο και στη γλώσσα που καταλαβαίνουν χρησιμοποιώντας ε, απλή γλώσσα και αποφεύγοντας την ε, υπερβολική νομική ορολογία που είναι δυσνόητη. Τώρα, άπαξ και έχει αρχίσει να ισχύει ο κανονισμό και τον έχουμε, και έχουμε αρχίσει να τον παρακολουθούμε, καταλαβαίνετε ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στο θέμα της συλλογή προσωπικών δεδομένων. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τους συνομοθέτες να πετύχουν τη σωστή ισορροπία κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου για όλα αυτά τα ζητήματα. Τέλος, γνωρίζουμε τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τη μετανάστευση και την εσωτερική ασφάλεια για το πακέτο αυτό όσον αφορά τη σνοριοφυλακή και την ακτοφυλακή. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, οι τελευταίες, και εφόσον εφαρμοστούν, η επεξεργασία των δεδομένων όσον αφορά επικό τρίτων χωρών, εδώ πρέπει να προσεχτεί όλος ιδιαίτερος. Δεν θα πρέπει όλους τους υπηκόους ε, τρίτων χωρών που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε σαν ενδυνάμει υπόπτους. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή σας που μας κάλεσε να έρθουμε και να παρουσιάσουμε τη δικιά μας άποψη όσον αφορά το τρέχον ζήτημα. Ευχαριστώ και την Επιτροπή και την Ολλανδική Προεδρία που αντάλλαξε μαζί μας πληροφορίες για το πώς προχωράει το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα περνάμε στους σκιώδες συζητητές. Έχουμε 15 συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο και θα φροντίσω να έχουμε αρκετό χρόνο για να συζητήσουμε αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα. Έχουμε χρόνο, αλλά προκειμένου να μπορέσουν όλοι να πάρουν το λόγο και μην ξεχνάμε ότι είναι και βράδυ στο Στρασβούργο, όλοι είμαστε κουρασμένοι, να είσαστε σύντομοι παρακαλώ, επί της ουσίας για να προλάβουμε και τα υπόλοιπα ζητήματα. Αρχίζουμε λοιπόν με τον ε, Πίτερ Νίλε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο. Να ευχαριστήσω πρώτα τον κύριο Πάμπριξ για την προθυμία του να συνεργαστεί και για την έκθεση αυτή. Και πρωτού μπω σε λεπτομέρειε, θα ήθελα να κάνω τρει γενικέ παρατηρήσει. Πρώτα απ' όλα η πολιτική μου παράταξη ε, έχει θετική άποψη για τη δημιουργία συνεροφυλακή και εκτοφυλακής ευρωπαϊκής. Δεν θα πρέπει να είναι αυστηρά ένα εργαλείο επιβολή νόμου αυτός ο οργανισμός πρέπει να έχει μια ολιστική προσέγγιση στην μετανάστευση. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η πρόταση τη Επιτροπή είναι πολύ φιλόδοξη. Από την άλλη, συντάχθηκε πάρα πολύ γρήγορα και ε, έχει έλλειψη αφήνει σε πολλά σημεία. Όσον αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόσο στον οργανισμό όσο και στη διαδικασία λήψη αποφάσεων, είναι πολύ περιθωριακός ο ρόλος αυτός. Ο στα θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών θα πρέπει το Κοινοβούλιο να έχει τον ρόλο ο οποίος τοποθετούνται από τις συνθήκες. Και άλλα έξι σημεία. Το πρώτο ήδη έχει αναφερθεί και είναι, το θέμα της κοινή ευθύνης. Η πρόταση της Επιτροπής δεν είναι καθόλου σαφής για το ποιος είναι υπεύθυνο για ποιο θέμα, πού και πότε η λογοδοσία του οργανισμού και των κρατών μελών είναι πολύ ασαφή σε πολλές περιπτώσεις όπως ε, τις επιστροφές, ε, την προστασία των δεδομένων κτλ. Θα ήθελα ο κύριος Πάμπριξ να μας παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια. Ένα δεύτερο σημείο αφορά τη μεγάλη βάση που δίνεται στις επιστροφές. Προβλέπεται ένα γραφείο επιστροφών που δεν θα βοηθάει μόνο τα κράτη-μέλη με τι επιχειρήσει επιστροφών, αλλά που θα τις ε, ε, δρομολογεί. Και το μήνυμα που δίνεται είναι ότι αυτό ο οργανισμό μπορεί να καταλήξει να είναι οργανισμό οργανισμός ε, επιστροφών. Ένα άλλο σημείο είναι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλώς όριζα τις προτάσεις της Επιτροπής. Όμως, όπως αναφέρθηκε ήδη, ανησυχώ για το ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για τις παραβιάσεις θεμελιδών δικαιωμάτων. Ένα επιπλέον σημείο είναι το σημείο των διασώσεων πολύ λίγα υπόθηκαν για τον ρόλο του νέου οργανισμού στις επιχείρησεις διάσωσης τη θάλασσα, ε, στο Αιγαίο και στα εξωτερικά σύνορα. Θα πρέπει να είναι μια προτεραιότητα ώστε να διασφαλιστεί ότι θα υπάρξουν ολοκληρωμένες ε, επιχειρήσεις διάσωσης και έγκαιρη παρέμβαση ώστε να αποφευχθούν ε, τέτοια θέματα. Αυτό είναι ένα πόσο στο κομμάτι της διαχείρισης των σύνορων και επίσης θα πρέπει να αποτελέσει και μία από τις αποστολές του οργανισμού. Και τώρα όσον αφορά την δομή του οργανισμού και τον ρόλο των θεσμικών οργάνων, ο ρόλος του εκτελεστικού διευθυντή είναι πολύ σημαντικός. Επίσης, ε, το Συμβούλιο του θα έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για ευαίσθητα θέματα. Και το Συμβούλιο προβλέπεται να έχει ένα σημαντικό ρόλο, όμως ε, το Ευρωκοινοβούλιο περιθωριοποιείται, γιατί αν ο εκτελεστικό διευθυντή έχει τόσο σημαντικό ρόλο, τότε θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει έναν πιο ισχυρό ρόλο και να μπορεί να διορίζει τον διευθυντή. Όσον αφορά τη διαφάνεια του προπολογισμού, σύμφωνα με την πρόταση τη Επιτροπή, έχει σημαντικό ρόλο το Ευρωκοινοβούλιο. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο προϋπολογισμός θα είναι λεπτομερής, ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς ποιο κομμάτι του προϋπολογισμού εξοδεύεται για επιστροφές, για επιχειρήσεις διάσωσης κτλ. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα ε, καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε και αυξημένη χρηματοδότηση για τον οργανισμό. Ευχαριστώ πολύ, Πίτερ. Η Χέλγκα Στίβεν, και από το ECR. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, εισηγητή. Είναι ένδειξη της καλής συνεργασία που είχαμε και που θα έχουμε και στο μέλλον. Είναι σαφές σε όλους μας ότι αυτός ο νέος κανονισμός είναι κάτι που θα πρέπει να έχει και ψηλή αλλά και να, ευθετηθεί, να εγκριθεί γρήγορα. Δεν θα ήθελα να ζήσουμε έναν ακόμα χρόνο γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ε, αυτό το εργαλείο ώστε να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς ε, τις καταστάσεις που θα αντιμετωπίσουμε τα το επόμενο χρόνο. Θα καταφέρουμε έτσι να ε, ενισχύσουμε την σωστή λειτουργία του Σέγγεν και γι' αυτό η ομάδα μας υποστηρίζει τον εισηγητή. Θα πρέπει να υπάρξει σωστή ισορροπία ανάμεσα στη Frontex και στα κράτη-μέλη και στην ε, παροχή ε, βοήθειας προς τα κράτη-μέλη από τη Frontex. Γι' αυτό υποστηρίζω ότι οι συστάσεις και οι παρεμβάσεις που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την χρήση της Frontex θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ειδική πλειοψηφία ε, στο Συμβούλιο. Η Frontex δεν θα ε, πρέπει να επιμένει ε, να βοηθήσει ένα κρατό μέλος, όμως θα πρέπει να υπάρχουν συνέπειε για τα κράτη-μέλη που θα αρνηθούν να δεχτούν τη βοήθεια από ένα άλλο μέλος με καταστροφικό τρόπο, με καταστροφικές συνέπειες. Γι' αυτό θα πρέπει να σε θέση το κράτος μέλος αυτό να κλείσει τα σύνορα. Θα πρέπει να υπάρχει συνέργεια μεταξύ των αρχών για να υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, αλλά παράλληλα να είναι και σαφής ο αντίκτυπος που θα υπάρχει στα, στους πόρους ε, για τα κράτη-μέλη, όπως είναι υπηρεσίες ε, επικοινωνίας, και άλλες δραστηριότητες. Βασικό στοιχείο είναι η ανάγκη να μοιραζόμαστε πληροφορίε. Θα πρέπει να μοιραζόμαστε πληροφορίε στα κρατημέλη μεταξύ μα όσον αφορά τι αδυναμίε, την τροτότητα ε, στα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτέ τι πληροφορίε θα πρέπει να μοιράζονται και από την Frontex. Είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να δίνουν πληροφορίε ε, στα σχετικά ευρωπαϊκά συστήματα. Ε, ο μηχανισμός παρακολούθησης και οι αξιολογήσεις ε, τροτότητας είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξεκινήσει να δημιουργεί πολιτικές ε, και να τις εφαρμόσει και όχι απλώς να αντιδρά στην κρίση. Μια κρίση που μπορεί να είναι και η κρίση του μέλλοντος. Είναι μια φιλόδοξη πρόταση δεν θα πρέπει για αυτόν τον λόγο να ε, παραβλέψουμε και το, την ομοθετική πτυχή. Να ευχαριστήσω και πάλι τον εισηγητή για το έργο του και ανυπομονώ να συνεργαστούμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ε, και τώρα, σκιώδης για την Άλτε, η Νάταλη Γκρίσπεκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μερικά λόγια να πω εν είδη εισαγωγής. Να εκφράσω τη θέση ομάδας μας δεν ταιριάζει απόλυτα με αυτά που είπε η συνάδελφος Έλκα. Να επενθυμίσω κάποια θεμελιώδη πράγματα. Όσον αφορά το χώρο του Σέγγεν, είμαι θα πεπισμένη, κάποιοι από μας ότι ο χώρος Σέγγεν δεν είναι βιώσιμος παρά μόνο αν τα εξωτερικά σύνορα προστατεύονται αποτελεσματικά. Και με πικρή ηρωνία διαπιστώνουμε αυτό το στοιχείο 30 χρόνια μετά τη δημιουργία του χώρου Σέγγεν. Είναι κάτι προφανές. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε την ελεύθερη διακίνηση των Ευρωπαίων. Ένα θεμελιώδες κεκτημένο. Ένα από τα πιο αρατά κεκτημένα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αν θέλουμε να διατηρήσουμε την Ευρώπη σαν χώρο άνευ εσωτερικών συνόρων, πρέπει προφανώς να ενισχύσουμε και να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα. Είναι ζωτική σημασία για την Ευρώπη και ζωτική σημασία πάνω απ' όλα για τους Ευρωπαίους. Όχι μόνο του οικονομικούς φορείς, αλλά του απλούς πολίτες που θέλουν να έχουν μια ενιαία ταυτότητα εντός της ποικιλομορφία των πολιτισμών. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειε απόψε. Είναι κοινή προσέγγιση αυτή. Σας σκιώδη για την ομάδα μου θέλω να υπογραμμίσω σχετικά με αυτό ότι προφανώς υποστηρίζουμε την πρόταση κανονισμού που αφορά τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος φυλάκων και ακτοφυλακή. θεωρούμε σαν ένα στάδιο, πρώτο στάδιο. Απαραίτητο. Και πάμε προς τον εξευρωπαϊσμό των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να ξεγελιόμαστε. Εδώ ακούμε, εδώ και μερικές εβδομάδες, κάποιους ηγέτες που αναφέρονται για την ακτοφυλακή αυτή, θεωρώντας ότι αυτή θα λύσει όλα τα προβλήματά μας όλα τα μεταναστευτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και τα εξωτερικά μας σύνορα. Είμαστε πολλοί και στην ομάδα μας που ζητήσαμε αναθεώρηση του συστήματος Frontex. Εδώ και πολλά χρόνια το ζητούμε. Θέλουμε να δοθούν αυξημένε αρμοδιότητες στη Frontex με τον ανάλογο προπολογισμό. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας γι' αυτό. Ζητούσαμε και τη δημιουργία πραγματικού ευρωπαϊκού σώματος θωριοφυλάκων. Εδώ και χρόνια το ζητούμε. Η πρόταση ακολουθεί σωστό δρόμο. Την υποστηρίζουμε. Εντάχει να αναφέρω κάποια πράγματα. Αυτή ε, η ομοσπονδιακή προσέγγιση πρώτη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια άμεση παρέμβαση σε περίπτωση απειλής για το χώρο Σέγγεν από όλα τα κράτη-μέλη θέλω να κατανοήσω καλύτερα πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τις αντιδράσεις κάποιων κρατών μελών όσον αφορά το μηχανισμό της προστασίας όλης της επικρατείας Σέγγεν. Δεύτερον, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Η πρόταση προτείνει τη δημιουργία ενός κέντρου αναλύσεως κινδύνου και συντάξεως εκθέσεων για τον κίνδυνο και αξιολόγηση του πόσο τροτάνε τα σύνορα των κρατών μελών κατάφερα τη διαφορά που υπάρχουν μεταξύ των δύο. Συνεχής έλεγχος της καταστάσεως, το ένα. Από την άλλη, θα χρησιμοποιεί το μηχανισμό στο άθρο 18 όταν χρειάζεται. Αυτοί οι δύο μηχανισμοί ίσως οδηγούν σε επικάλυψη προσπαθειών. Μήπως θα έπρεπε να έχουμε ένα και μοναδικό κέντρο που σε πραγματικό χρόνο θα διαπιστώνει ποια είναι η κατάσταση. Τρίτον, ε, χαιρετίζω το έργο το αποτελεσματικότατο της Την προσπάθεια συντονισμού, συμφιλιώσεως των απόψεων. Συμφωνώ με τον εισηγητή, πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Όμως, Μήπως ε, αν καταργήσουμε το Εποπτικό Συμβούλιο είναι κακό. Χρειάζεται να υπάρχει ισορροπία δυνάμεων στο φορέα. Μήπως δημιουργείται κίνδυνος έτσι. Το αντίθετο της επικάλυψης που ανέφερα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι σε αυτό. Υπάρχουν σημαντικότατα σημεία που εκκρεμούν. χρειάζονται διευκρίνηση. Το θέμα της διάσωσης, ανθρωπιστική πτυχή. Αυτό το γραφείο επιστροφή, αν θέλετε, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων μετά. Τα βασικά στοιχεία αναφέρθηκαν σαφέστατα προηγουμένω. από την ομάδα του οργανισμού. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η Σκά Κέλλερ που είναι η συγγήτρια για τους πράσινους έχει το λόγο. Η σκιώδη συγγήτρια. Ευχαριστώ. Θέλετε να μιλήσετε πρώτοι? Λέει Σκά. Λυπάμαι, λυπάμαι, λέει ο Πρόεδρος. Συγγνώμη, κουράστηκα. Έτσι μου το γράψανε. Το βλέπετε και στην ημερήσια διάταξη. Αυτή τη σειρά ακολουθείτε. Ζητώ δύο φορές συγγνώμη. Και εγώ δεν πρέπει να κατηγορώ τη Η Μαρίνα Άλμπεο για την ομάδα της ΚΟΕ και ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς η ομάδα μου ποτέ δεν αγάπησε τη Frontex γιατί ο ρόλος της δεν είναι να σώζει ζωές, κάθε άλλο μην το ξεχνάμε. Είναι ένας οργανισμός για τον έλεγχο των συνόρων, για να προστατεύει τα σύνορα, και άρα τον μετανάστη τον βλέπει σαν εχθρό. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο της Ευρώπης οχυρού και θεωρεί εγκληματική ενέργεια τη μετανάστευση. Οπότε η πρόταση αυτή τι κάνει, κάνει τη Frontex ένα εργαλείο ακόμα πιο απάνθρωπο και με ακόμα λιγότερες εγγύσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σήμερα βλέπουμε τις συνέπειες του μοντέλου αυτού της Ευρώπης οχυρού, της Ευρώπης των ε, τυχών. Είδαμε τι έκανε η Frontex μέχρι τώρα. Είναι αυτή η πραγματικότητα. Συνεπώς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση σαν να μην περίμεναν χιλιάδες την ειδωμένη οι οποίοι ζουν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, εγκλωβισμένοι. Έχουμε χιλιάδες νεκρούς στη Μεσόγειο. Έχουμε τόσους μετανάστες και μετανάστρες εγκλωβισμένους και ανθρώπους οι οποίοι με τη βία μεταφέρονται. Αυτό είναι το μοντέλο της Ευρώπης οχυρού και αυτό ακριβώς αντικατοπτρίζει και η Frontex. Σήμερα όμω δεν χρειαζόμαστε περισσότερου ελέγχου σύνορων, δεν χρειαζόμαστε περισσότερου αστυνομικού στα σύνορα, δεν χρειαζόμαστε περισσότερη εξωτερήκευση των σύνορων ώστε χώρε όπω η Τουρκία να κάνουν του δεσμοφύλακε. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα δεν είναι περισσότερη Frontex, ούτε την παλιά ούτε την καινούρια. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι δρόμους νόμιμους, ώστε να μην χρειάζεται κανείς να κινδυνεύει τη ζωή του στη θάλασσα. Η διεθνής νομιμότητα να τηρηθεί, αυτό θέλουμε, και να τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εγώ αυτό δεν το βλέπω σε αυτή την πρόταση που εξετάζουμε σήμερα. Δεν καταλαβαίνω. Οι πληροφορίες για τα δικαιώματά τους και η διαδικασία προσφυγής είναι πράγματα τα οποία θα λέμε στους ανθρώπους αυτούς όταν είναι στη θάλασσα, όταν φτάνουν ε, στις ακτές μας ή όταν τους επιστρέφουμε στην Τουρκία. Δεν έχω καταλάβει πότε θα τους ενημερώνουμε για τα δικαιώματά τους όπως λέτε. Στην πρόταση αυτή αυτό που κάνουμε είναι να αντιμετωπίζουμε τους μετανάστες σαν να είναι εγκληματίες. Όλο το κείμενο της πρότασης αυτό κάνει. Συνδέει τη μετανάστευση με την έλλειψη ασφάλειας και από όσου μιλήσαν εδώ αυτό κάνανε. Συνδέανε τη μετανάστευση με την τρομοκρατία. Άρα για να διατηρήσουμε την ασφάλεια μέσα στο χώρο Σέγγεν πρέπει να προστατευτούμε, να προστατεύσουμε τα σύνορά μας. Από ποιον. Μα δεν είναι εχθροί. Αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να βρουν ένα μέλλον για τα παιδιά τους. Είναι σαν να ακούω την άκρα δεξιά. Αυτοί που συνέταξαν δηλαδή την πρόταση αυτή, αυτό μου θυμίζουν για τον κανονισμό της Frontex. Εμείς λοιπόν από την ομάδα μου, την QE NLG, δεν συμμεριζόμαστε ούτε τους στόχους, ούτε την αναγκαιότητα, ούτε το πνεύμα της πρότασης αυτής για την νέα υπηρεσία Frontex. Από πλευρά του Συμβουλίου φαίνεται σα πρότεινα να αλλάξετε όνομα της πρότασης. Την πρόταση θα μπορούσατε να την πείτε υπηρεσία για την επιστροφή, υπηρεσία για τις διαβίες επιστροφέ, χιλιάδων ανθρώπων. Και σα υπενθυμίζω ότι αυτή η με μεταφορά των ατόμων αποτελούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητα. Νομίζω λοιπόν ότι κάτω από αυτούς τους όρους εμείς θα υποβάλουμε τις τροπολογίες μας που βέβαια θα είναι μια τροποποίηση της συνολικής πρότασης, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Η πράσινη τώρα, Σκά έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για την πρότασή του και ευχαριστώ όλους τους προλαλήσαντες. Έχω μία-δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο άρθρο 26 παραδείγματος χάρη 2β αναφέρεστε στο εξή ότι η Frontex θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες προς τα κράτη-μέλη πληροφορίες όσον αφορά τις τρίτες χώρες επιστροφής δεν είναι ξεκάθαρο τι είδους πληροφορίες θα παρέχονται πληροφορίες για τη γενική κατάσταση η ΆΣΟ κάνει εκθέσεις κατά χώρα τι είδους πληροφορίες εννοείται μετά αναφέρεστε στον χώρο των χώρων υποδοχής, hotspot. Είναι διαφορετικό το hotspot area από το hotspot. Είναι περιοχή του hotspot, είναι ταυτόσιμο με το hotspot. αυτή είναι δύο συγκεκριμένε ερωτήσει που απευθύνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σαν πράσινοι θα υποβάλουμε μερικές τροπολογίες παρόλο που κάποια από τα ζητήματα που συζητήσαμε του Σκιώδης ήδη αντικατοπτρίζονται στην έκθεση του εισηγητού και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Όσον αφορά θεμελιώδη δικαιώματα, είναι σημαντικό να ενισχύσουμε το ρόλο της έρευνας και διάσωσης. Τον ανέφεραν και συνάδελφοι. Είναι σημαντικό και για τις δραστηριότητες ακτοφυλακής. Η λογοδοσία στο Κοινοβούλιο, που τον έφεραν και αυτό συνάδελφοι. Αυξημένο ρόλο του Κοινοβουλίου όσον αφορά την επιλογή του εκτελεστικού διευθυντού. Αν αυτό το άτομο, εκείνο ή εκείνη έχουν περισσότερη εξουσία, θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυτά που προβλέπουμε και για άλλες υπηρεσίες, για άλλους οργανισμούς. Κάτι άλλο σημαντικό. Να μην επιτρέψουμε τις επιστροφές από τρίτες χώρες. Έχουμε επιστροφές σε τρίτε χώρε. Αν η Frontex θα κάνει επιστροφέ από τρίτε χώρε. Δηλαδή άνθρωποι που είναι σε τρίτες χώρες και επιστρέφονται σε τέταρτη, σε μια άλλη χώρα. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Δηλαδή κατά πόσο γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα αν σεβόμαστε την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Και τα δικαιώματά του υποβάλλουμε, η τροπολογία όσον αφορά την ευθύνη και τη ε, λογοδοσία στην Frontex. Δεν είναι σαφές ποιος είναι υπεύθυνο γιατί. Όσον αφορά την ε, υποβολή ενστάσεων θα υποβάλουμε ε, τροπολογίες για να αφιγραμμιστούμε με την έκθεση την οποία συνέταξα με την Ρομπέρτα Ματσόλα. Από τη στιγμή που θα έχουμε θέση του Κοινοβουλίου θα πρέπει όλο το θέμα να το αντιμετωπίσουμε σφαιρικά για τη Frontex. Θα υποβάλουμε τροπολογίες για τις δυνατότητες παρέμβασης της Frontex παρά τη βούληση των κρατών μελών. Ενάντια στη βούληση των κρατών μελών. Κάτι που προανέφερα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να λάβουμε υπόψη του Ευρωπαϊκού Κέντρου, του EDPS μάλλον. δεν είχαμε δυνατότητα να ακούσουμε την άποψή τους πριν υποβάλει την Προτασία της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα πολύτιμα σχόλιά τους και δύο ερωτήσεις, πιο αόριστες ίσως αυτές. Αναφέρεται ότι η Frontex έχει σαν καθήκον να εξασφαλίζει την εσωτερική ασφάλεια. απευθύνω ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κύριο Λετζέρη. Στα σύνορα γίνονται έλεγχοι. Ποιος εισέρχεται. Αν επιτρέπεται λαθρεμπόριο όπλων, αν μπαίνουν όπλα ή όχι. Αυτό είναι ένα κομμάτι της εσωτερικής ασφαλείας, αλλά τα σύνορα δεν είναι αποκλειστικά το αποκλειστικό στοιχείο της εσωτερικής ασφαλείας. Πώς γίνεται αντιληπτό αυτό αν μπει στα καθήκοντα της Frontex αυτό, δηλαδή στην υπηρεσία των έλεγχων των συνόρων αναθέτης καθήκων ε, φύλαξης και ε, διαφύλαξης εσωτερικής ασφαλείας. Το θέμα του προπολογισμού αναφέρθηκε. αυτό θα έχει συνέπειες. Αν η Frontex έχει νέες αρμοδιότητες, υπάρχουν συνέπειες. Και αν όλα όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνουν, τότε ποιες θα είναι οι οικονομικές ανάγκες της ε, Frontex θα μπορούσατε να μας δώσετε περίπου κάποιο αριθμητικό στοιχείο για το ποσό που απαιτείτε. Ευχαριστώ. Η ευθυντή δεν είναι εδώ ο κύριος Καράς. Αλλά παρακαλώ εσείς θα μιλήσετε εκ μέρους του. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ για τις πληροφορίες, πολλές πληροφορίες πράγματι όσον αφορά το νέο αυτό οργανισμό για την προστασία των εξωτερικών αλλά και εσωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ όταν ολόκληρο το σύστημα φαίνεται να καταραίει, το σημερινό Frontex έχει ως στόχο να προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα. Αλλά δεν έγινε αυτό. Αυτό που έκανε ήταν να ψάχνει στη θάλασσα και να διασώζει. Οπότε, η νέα αυτή υπηρεσία, αυτός ο οργανισμός θα ελέγχει τα εξωτερικά σύνορα και κυρίως τα θαλάσσια σύνορα. Εγώ θέλω να ξέρω όμως τι θα κάνει αυτά τα θαλάσσια σύνορα εκτός από το να ψάχνει και να σώζει ζωές. Ακούσαμε επίσης ότι δεν θα πληγεί η εθνική κυριαρχία. Μα πώς, θα πληγεί. Γιατί ο οργανισμός αυτός έχει το δικαίωμα να δρά και να αναπτύσσεται στη εθνική επικράτεια εάν κρίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι χρειάζεται να παρέμβει. Πώς και ποιος θα το αποφασίζει αν υπάρχει κάποια δυναμία σε μια χώρα και πρέπει να αναπτυχθούν οι δυνάμεις του. Με άλλα λόγια, πρακτικά μιλώντας αλλά και οικονομικά μιλώντας, πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό. Στη Σουηδία θέλουμε να επιστρέψουν 80.000 ανθρώπους τα επόμενα δύο χρόνια. Θα μπορεί αυτός ο οργανισμός να βοηθήσει οικονομικά, πρακτικά. Και αυτό είναι κάτι που θέλω να ρωτήσω. Αλλά πάνω απ' όλα νομίζω <coughs> ότι οι χώρες μέλη πρέπει να ελέγχουν τα δικά τους σύνορα και νομίζω ότι η σημερινή Frontex πρέπει να είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των εξωτερικών σύνορων. Ευχαριστώ από το ΙΕΝΕΦ, ο κύριος Λιμπρέτο τώρα, τελευταίος από τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πάπριξ, ο οποίος πολύ καλά ηγήθηκε των εργασιών μας. Το κείμενο αυτό έχει να κάνει με μια μεταναστευτική κρίση χωρίς προηγούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Frontex δεν μπόρεσε να την αντιμετωπίσει είναι η απόδειξη της ανεπάρκειάς της. Και τώρα θέλουμε να την αντικαταστήσουμε από έναν άλλον οργανισμό συνοριοφυλακής και εκτοφυλακής. Το αρχικό κείμενο ήταν πολύ ανησυχητικό όσον αφορά την εθνική κυριαρχία των χωρών μελών. Χάρη στη δουλειά που έγινε όμως με επικεφαλή στον κύριο Πάμπριξ βελτιώθηκε κάπως το κείμενο. Για παράδειγμα βγήκε το Εποπτικό Συμβούλιο ε, του οργανισμού. Άρα θα έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία, τόσο το καλύτερο. Διαπιστώνω επίσης ότι επιμείναμε πολύ προκειμένου να βοηθάει ο οργανισμός της χώρες και όχι ανταγωνιστικά να λειτουργεί. Αναφέρεται όρος assistance στα γαλλικά, ε, βοήθεια, που είναι μια λέξη που δηλώνει ταπεινότητα. Καλό λοιπόν και αυτό. Επίσης διαπιστώνω ότι με περισσότερη σαφήνεια αναφέρεται τώρα ότι λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ο νέος αυτός οργανισμός. Επίσης ότι η αξιολόγηση του πόσο τροτή ευάλωτη είναι η κάθε χώρα και τα σύνορά της, επίσης είναι κάτι που θα υποβάλλεται σε αυτούς τους δύο θεσμούς. Ε, κατά τα άλλα, πια δεν θα είναι σε όλες τις χώρες για να λειτουργούν σαν κατάσκοποι, επιτρέψτε μου να το πω έτσι, αλλά μόνο στις χώρες που έχουν εξωτερικά σύνορα. Κάτι είναι και αυτό. Παρόλο που δεν φτάνει, γιατί πλήττει σε μεγάλο βαθμό την κυριαρχία, την εθνική κυριαρχία, το κείμενο αυτό. Επαναλαμβάνω ότι θα πρόκειται για άτομα του οργανισμού αυτού που θα πηγαίνουν και θα λειτουργούν ως κατάσκοποι στις χώρες μέλη. Για μένα όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Άπαξ και μια χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα, είναι θεμητό να το συζητήσει με τις γείτονες χώρες, να προσπαθήσουν να βρούνε κοινέ λύσεις μεταξύ τους. Αλλά έτσι να βάζουμε σε κυδαιμονία μια χώρα μέλη, ε, μέλος, κατά τη γνώμη μου αυτό είναι απαράδεκτο. Εξάλλου μπορεί να καταλήξει σε συγκεκριμένες αποφάσεις του εκτελεστικού διευθυντή που θα ζητήσει από τη χώρα μέλος να πάρει διορθωτικά μέτρα. Κάτι άλλο που θεωρώ απαράδεκτο είναι η ομάδα αυτή ταχείας αντίδρασης που είναι στη διάθεση του οργανισμού. Πάλι εγώ βλέπω ότι χρησιμοποιούμε κεντρικά τους σπόρους και δεν θα έπρεπε. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να φανταστούμε μία χώρα να πηγαίνει να βοηθά μία άλλη εφόσον τη το ζητήσει, αλλά όχι έτσι κεντρικά να υπάρχει αυτή η εφεδρεία κεντρικά. Και έρχομαι και στο χειρότερο άρθρο που είναι το άρθρο 18 που αναφέρεται στη ταχεία αντίδραση και που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνει έτσι αυταρχικά άπαξ και μια χώρα έχει την ατυχία να μην έχει πάρει τα διορθωτικά μέτρα τα οποία συστήνει ο οργανισμός. Αλλά και εδώ υπάρχει κάποια βελτίωση χάρη στον κύριο Πάμπριξ. Στην αρχή ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκείνη η οποία αποφάσισε και με εκτελεστικές πράξεις προχωρούσε. Τώρα βελτιώνεται η κατάσταση. Είναι το Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία. Παρ' όλα αυτά πλήττεται η εθνική κυριαρχία και για μένα είναι απαράδεκτο, όπως επίσης και για την ομάδα μου. Και τελειώνω με κάτι πιο γενικό. Ο 21ος ε, αιώνας βλέπει τα έθνη να επανέρχονται με όλη τους τη δόξα. Το κείμενο όμως αυτό δεν λαμβάνει υπόψη αυτό το ιστορικό γεγονός θα ενισχύσει τον ευρωσκεπτικισμό στις διάφορες χώρες μέλη. Πρόσφατα το είδαμε με το δημοψήφισμα στις κάτω χώρες. Όπου να είναι θα έχουμε και ένα άλλο με το Brexit. Και διαπιστώνω ότι παντού αυτό που ονομάζετε εσείς λαϊκισμός ανεβαίνει και ουσιαστικά δεν πρόκειται για λαϊκισμό, αλλά πρόκειται για εθνική κυριαρχία. Ευχαριστώ που περιμένετε τόσο πονητικά. Σας παρακαλώ να μιλήσετε μόνο για δύο λεπτά, ώστε να έχουμε χρόνο στη συνέχεια να δώσουμε και πάλι το λόγο στην Επιτροπή και στην Προεδρία και στη Frontex, όμως και στον εισηγητή. Σας παρακαλώ λοιπόν να περιοριστείτε, σε δύο λεπτά. Κύριε Κοέγιο, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που αντιδράσαμε γρήγορα, γιατί όντω επήγει το θέμα και θα έπρεπε να αντιδράσουμε έτσι γρήγορα. Όπως το είπαν και άλλοι πριν από μένα, πρέπει να πω και εγώ ότι το κείμενο αυτό δεν είναι πανά και δεν λύνει όλα μας τα προβλήματα, πρέπει να πάρουμε και άλλα μέτρα. Κάποιες παρατηρήσεις όμως έχω να κάνω. Πρώτον, όσον αφορά το εξή που θέλω να υπογραμμίσω. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στην αξιολόγηση του νέου συστήματος Σέγγεν και του νέου συστήματος που αξιολογεί το ευάλωτο ή το τροτό των συνόρων μιας χώρας. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ένα και στο άλλο. Θέλω να ξέρω λοιπόν ποιο είναι το εύρος εφαρμογής της μιας και της άλλης περίπτωσης και πώς συμπληρώνει το ένα σύστημα το άλλο. Εγώ νομίζω ότι όταν πρόκειται για την αξιολόγηση του τρότου, του ευάλωτου, εδώ πρέπει να υπογραμμίζουμε το εξή. Ο νέος οργανισμός θα είναι αυτός που θα το χειρίζεται. Με το σύστημα Σέγγεν υπήρχαν αδυναμίες που είχαμε καταγγείλει, αλλά δεν τις παρούσε. Έπειτα όσον αφορά τον αποκλεισμό από το χώρο Σέγγεν μιας χώρας. Προβλέπεται, αλλά είναι πάρα πολύ περιορισμένο. Το γεγονός ότι το βρίσκουμε και πάλι σε αυτήν εδώ την πρόταση, δεν καταλαβαίνω. Δεν θα πρέπει ο κανονισμός να χρησιμεύει για να παρακάμπτεται ένας μηχανισμός που ήδη υπάρχει και που βρίσκεται σε μια διαφορετική νομική πράξη. Επόμενη παρατήρηση οι συνοριοφύλακες στο μέλλον θα έχουν πιο ενεργό ρόλο όσον αφορά τις επιστροφές. Μια αξιόπιστη πολιτική επιστροφών είναι η άλλη πλευρά του νομίσματος, μια δηλαδή γενναιόδορης πολιτικής ε, ασύλου. Πάνε μαζί αυτά τα δύο. Πρόεδρε, θέλω να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής στο εξής. Πρέπει ξεκάθαρα να λέμε ο διοργανισμός αυτός πρέπει να συνδέεται με τον κανονισμό 656 του 2014 που ορίζει τους κανόνες για μέτρα ελέγχου στα πλαίσια λειτουργίας της Frontex και όσον αφορά τις έρευνες στη θάλασσα και τη διάσωση. Η εφαρμογή του κανονισμού λοιπόν 656-2014 για μένα πρέπει να γίνεται αυτόματα. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μια διαφορετική ερμηνεία από αυτήν, τότε πρέπει να το συμπεριλάβει στον κανονισμό για να πει ξεκάθαρα ότι ο οργανισμός λειτουργεί διαφορετικά. Αλλιώ πρέπει να λέει ρητά ότι δεσμεύεται από τον κανονισμό αυτόν. Ευχαριστώ, Κλοντ. Είναι αφιλεγόμενο το θέμα. Όλοι θεωρούμε ότι αυτό χρειάζεται η εφαρμογή του ΣΕΝ η διαφύλαξη των συνόρων, ότι θα πρέπει να δώσουμε μια λύση σε αυτή την κρίση. Όμως από την άλλη πλευρά δεν έχουμε ακόμα μια κοινή θέση για την πολιτική ασύλου. Και γι' αυτό βλέπω ότι δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα για αυτό το νέο σύστημα, χωρίς να ξέρουμε τι είδου πολιτική θα αναπτύξουμε. Και συμφωνώ απόλυτα ότι είναι η δίωξη του ίδιου νομίσματο. να καταλάβουμε τι είναι μια νέα μορφή τι είναι τέλο πάντων. επίση το πεδίο εφαρμογή ε, δεν είναι σαφές, δεν ορίζεται. Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογή, γιατί μια μόνιμη ακτοφυλακή γνωρίζουμε ήδη ότι σε κάθε κάποιος μέλος έχει διαφορετική λειτουργία. Αφορά αυτή τη μεταναστευτική πίεση και πώ την αντιμετωπίσουμε ή αφορά και άλλες ε, ε δραστηριότητες που έχουν εκτοφυλακές. Και βλέποντας τα ευρωπαϊκά σύνορα είναι διαφορετικό αν δούμε τα σύνορα με τη Ρωσία ή τα σύνορα της Μεσογείου είναι διαφορετικά τα προβλήματα από διαφορετικές λύσεις. Φανταστείτε λοιπόν ήταν υπουργό άμυνα κ. Παμπρίξ τη Λετωνία. Επομένω, καταλαβαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθούν ε, κάποιο είδος ευρυδικών προσφύγων, ε, οικολογικών προσφύγων. Επομένω, αυτό το νέο επιχειρησικό ε, σύστημα θα αφορά και τέτοιου είδου περιπτώσει ή όχι. Θα πρέπει επομένω να είμαστε πολύ σαφείς για να ξέρουμε ότι αφορά άμεσες απειλές. Γιατί η συνεργασία με τον Νότο είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Άρα πρέπει να έχουμε ένα ξεκάθαρο παιδί εφαρμογή, σαφή λειτουργία, μια συστημική θεώρηση σε σχέση και με την πολιτική ασύλου. Επίσης, θα πρέπει να δούμε τι χρειάζεται για να ενισχύσουμε τα σύνορα. Χρειάζονται τεχνικές λύσεις πέρα από το προσωπικό και το βλέπουμε αυτό και στην Ελλάδα και οπουδήποτε, ε, οπουδήποτε συστήματα καταγραφής και άλλα τεχνικά συστήματα και τέλος προστασία δεδομένων φυσικά. Με όλο το σεβασμό στις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ξέρουμε ποια είδη δεδομένων χρειαζόμαστε και γιατί και για τη μετανάστευση δεν κάνουμε λόγο μόνο για δεδομένα που χρησιμοποιούμε μόνο για τρεις μήνες, αλλά που θα χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον, που θα πρέπει να τα επανασυλλέξουμε. Και θα πρέπει να ξέρουμε ποια θα είναι η βάση δεδομένων που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε για να έχουμε μια αποτελεσματική πολιτική. Είναι πολύ αργή διαδικασία όμως χρειάζονται τα δεδομένα για την, επανεγκατα... για την ε, μετεγκατάσταση και γι' αυτό θα πρέπει να τα στήσουμε όλα αυτά ξεχωριστά. Υπάρχουν πολλές ασάφειες λοιπόν. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε έτοιμοι για να βρούμε κάποια κοινή λύση. Μαρή Κριστίν Βέρτζια, παρακαλώ. Εγώ θεωρώ ότι σε αυτό την Επιτροπή γίνονται συζητήσεις όλο και πιο σουραλιστικές. Ακούμε να λένε ότι όλα αυτά που ακολουθούν περισσότερη Ευρώπη είναι καλά και στο ίδιο κείμενο έχουμε άλλους που λένε ότι είναι δραματική κατάσταση και παρεμποδίζεται εξουσία των κρατών μελών. Το θέμα είναι το κείμενο, στο, σύμφωνο το κείμενο ποιος κάνει τι. Όλοι γνωρίζουμε τα κράτη-μέλη θέλουν να διαφυλάσσουν τις αρμοδιότητές τους όταν θέλουμε να προωθήσουμε κυρίως τα θεμελιώδη δικαιώματα. Κυρίως όμως όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, όταν υπάρχει πρόβλημα τρομοκρατίας, φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έκανε τη δουλειά της. Το είδαμε και με τα δεδομένα των επιβατών. Η Γαλλίδα, ξέρω τι έγινε στη Γαλλία. Δεν ε, θα είχε εμποδίσει τις επιθέσεις στο Παρίσι η ανταλλαγή δεδομένων επιβατών. Έχουμε πρόβλημα στα σύνορα, φαίνεται κρίση μεταναστών. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτόν τον όρο, θα επανέλθω. Ναι, αλλά ποιο ελέγχει σήμερα τα σύνορα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη-μέλη τη. Πού είναι τα ανθρώπινα μέσα, τα οικονομικά μέσα, 13 δισεκατομμύρια από το 2000 για την προστασία των συνόρων. Ναι, αλλά θα έπρεπε να ελέγχουμε τη χρήση των χρημάτων αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον έλεγχο των συνόρων που δεν κάνουν οι χώρες μέλη. Οπότε αναρωτιέμαι, τι συζητάμε εδώ. Και αν πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα, είναι πράγματι για να αποφύγουμε ο μετανάστης, ο πρόσφυγας, γιατί κυρίως έχουμε να κάνουμε με προσφυγική κρίση. 60 εκατομμύρια μετατοπισμένοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεπεραστεί 0,2% του πληθυσμού της. Μα τι κάνουμε περπατάμε με το κεφάλι κάτω και τα πόδια πάνω και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να ελέγξει τι κάνουν οι χώρες μέλη, αν ελέγχουν όντως τα σύνορα, τα εξωτερικά ή όχι. Μα αν τηρούσαν όλοι το διεθνές δίκαιο για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων, τότε θα πηγαίναμε μπροστά ενώ τώρα προσπαθούμε να κάνουμε άλματα με κάτι καινούριο που δεν θα λύσει απολύτως τίποτα. Κριστίν Λαμπρά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, όσα ακούσαμε δεν θα τα επαναλάβω, αλλά συμφωνώ για τα σημεία που εμείς σοσιαλιστές προβάλλουμε. Θέλω να επανέλθω όμως σε κάτι για το οποίο μίλησα πολλές φορές στην Επιτροπή μας και είναι σημαντικό να υποβάλουμε τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση γιατί δεν τις βλέπω προς το παρόν. Πρόκειται για τη συνεργασία με τρίτες χώρες και με συμφωνίες εργασίες. Το άρθρο 53 του σχεδίου κανονισμού λέει ότι ο νέος οργανισμός θα μπορεί να συνεργαστεί με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών στα πλαίσια συμφωνιών εργασίας όπως ισχύει τώρα με την Frontex. Έτσι προβλέπεται να προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και από τις δύο πλευρές και των ετούντων άσυλων, αλλά είναι κάτι για το οποίο δεν μπορούμε να υποελευθεύσουμε τίποτα και ούτε είναι δεσμευτική η δέσμευση αυτή. Όπως και ο Πίτερ το είπε πριν από λίγο και για αυτό το θέμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορεί να ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο στα πλαίσια των συμφωνίων αυτών. Θα πρέπει να ενημερώνεται πριν συνεχθούν αυτέ οι συμφωνίε και τακτικά για το τι περιλαμβάνουν. Και ο οργανισμό θα πρέπει ετησίω να υποβάλει έκθεση προ αυτή την κατεύθυνση. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι μόνο η Επιτροπή που πρέπει να εγκρίνει τι συμφωνίε αυτέ, αλλά και το Κοινοβούλιο. Να ενισχυθεί διαφάνεια λοιπόν και να υπάρξει δημοκρατικό έλεγχο είναι κάτι που εφαρμόζεται και όσον αφορά τα δημοσιονομικά για την τεχνική αρρωγή. Έπειτα, η επεξεργασία πρόσφυγων που προβλέπει το άρθρο 72 του κανονισμού περιλαμβάνεται και στις συμφωνίες εργασίας και στις συμφωνίες που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο, στις συστάσεις μάλλον, του συνήγορου του πολίτη δεν πρέπει όλα αυτά να είναι συμβολικά, μόνο στα χαρτιά. Όντω πρέπει να λαμβάνετε δράση, άπαξ και υπάρχει παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι παρατηρητέ τρίτων χωρών που προσκλήθηκαν από τον οργανισμό να συμμετάσχουν σε δράσει στα εξωτερικά σύνορα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και επίση να ληφθεί υπόψη το άρθρο 35 που αναφέρεται στην κατάρτιση των συνοριοφυλάκων, ακτοφυλάκων και άλλων ε, φορέων των χωρών μελών προκειμένου να μπορούν να εντοπίσουν και να ασχοληθούν με τα πιο ευάλωτα άτομα κυρίως εκείνα που είναι θύματα ελαφρεμπορίου λευκής σαρκός. Ευχαριστώ. Άννα Γκόμες, παρακαλώ. Ε, έγραψα μια έκθεση πριν από κάποια χρόνια για την ασφαλεία στη θάλασσα και με εντυπωσιάζει τώρα ε, η ακτοφυλακή που ε, ουσιαστικά περιλαμβάνει στρατιωτικέ επιχειρήσει, δραστηριότητε. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έχουμε τράφικινγκ στα σύνορα. τα σύνορα, ναι, αλλά δεν αναφέρεται τίποτα γι' αυτό. Έχουμε τεράστιο πρόγρα... πρόβλημα. Δεν αναφέρεται πουθενά. Η μόλυνση, ούτε σε αυτήν την αναφορά. υποδομές. Ούτε σε αυτό γίνεται αναφορά. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να απελάβνουμε ανθρώπους, πρόσφυγες και μετανάστες και συμφωνώ με την ΚΟΕ. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι ένας μηχανισμός απέλασης. Ούτε έρευνες, ούτε επιχειρήσεις διάσωσης. Δεν είναι αυτά οι στόχοι και παρόλο που έχουμε ήδη μια επιχείρηση που λαμβάνει χώρα που έχει σώσει 9.000 ζωές Σοφία, Σοφία η οποία διεξάγεται υπό διεθνή νομοθεσία και αποτελεί ένα κεντρικό ουσιαστικό στοιχείο αυτής της αποστολής. Αυτό είναι πολύ λιγότερο από την ε, επιχείρηση Σοφία που εφαρμόζεται, που παρά τα σωστά επιτεύγματα, τη διάσωση ζώων, έχει κάποια όρια. Γιατί οι παράνομοι διακινητές καλούν ουσιαστικά άτομα από την επιχείρηση Σοφία για να διασώσουν τους πρόσφυγες. Είναι υπέρ της εκτοφυλακής λοιπόν, αλλά όχι όπως προτείνεται. Όχι με αυτά τα χαρακτηριστικά και ειδικά σε μια εποχή, σε έναν καιρούς όπου υπάρχει αυτή η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για την οποία είμαι πεπισμένη ότι δεν είναι απλά ανήθικη, αλλά και καθόλου πρακτική μετά από τι επισκέψει που έκανα στην Ελλάδα πριν από δύο εβδομάδε. Όσον αφορά τη διάθεση του Σέγγεν, βλέπω την Επιτροπή ή το Συμβούλιο να δείχνουν το δάχτυλο στις χώρες αυτές που κατήργησαν ουσιαστικά, καταστρατήγησαν το Σέγγεν. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, ας μην γελιόμαστε. Πρέπει να ντρεπόμαστε. Υπέρ της εκτοφυλαϊκής, αλλά όχι όπως προτείνεται. Είναι ένας μηχανισμός απέλασης, έτσι όπως προτείνεται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας πω εγώ τι έχω κατάλαβει από όλα αυτά και από την έκθεση. Έχουμε μια κατάσταση που πρέπει να έχουμε ε, ισχυρό έλεγχο των εξωτερικών συνόρων μας. Κάποια κράτη-μέλη αισθάνονται πίση και δυσκολεύονται να παρέχουν αυτό τον έλεγχο και αυτό είναι ένα εργαλείο αλληλεγγύης ώστε από κοινού ε, να συνεχίσει η Frontex ε, να κάνει τις έρευνες, τις διασώσεις, να εντοπίσει τους παράνομους διακινητές, τους τράφικερς κτλ με περισσότερα μέσα, με, μεγαλύτερη δύναμη και παράλληλα να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη που πρέπει να ελέγξουν τα εξωτερικά του σύνορα. Αυτό κατανοώ εγώ και συμφωνώ με τη συνάδελφο ότι πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια. Και γι' αυτό το λόγο ε, επικροτούμε την πρόταση του κυρίου Πάμπριξ γιατί έχει σαφήνεια και όσον αφορά τώρα τον πυρήνα του θέματος η διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας θα υπάρξει με τη βοήθεια των θεσμικών οργάνων και μπορούμε να βρούμε αυτή την ισορροπία γιατί έχουμε από τη μία την ειδική πλειοψηφία όπως την Επιτροπή στο Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη από την άλλη θα πρέπει να συμφωνούν ε, για την προτινόμενη επιχείρηση και δεν θα τους επιβάλλεται μια επιχείρηση. Αυτό κατάλαβα εγώ. Εκεί που θα ήθελα περισσότερη σαφήνεια από τον εισηγητή ένα πιο δύσκολο σημείο για μένα είναι όταν ένα κράτος μέλος δεν είναι ικανό να ε, εξασφαλίσει επαρκή έλεγχο και δεν ε, ακούει τις συστάσεις το αν θα πρέπει ένα άλλο κράτος μέλος, τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να ε, παρισάγουν εσωτερικό συνορικό έλεγχο για έξι μήνες. Θα υπάρχει δυνατότητα αυτή να υπάρξει και πάλι έλεγχος από μια χώρα στα εσωτερικά σύνορα, άμα μια χώρα στα εξωτερικά σύνορα δεν μπορεί να εξασφαλίσει τον ε, έλεγχο. Και επίση Frontex θα βοηθήσει τα κρατημέλη στι επιστροφές, χωρίς όμως ε, να αφαιρέσει την αρμοδιότητα για τι επιστροφές από τα κράτη-μέλη. Επίσης θα ήταν πολύ σημαντικό να υπάρξει ένας εξωματούχος για ε, ε, την διασφάλιση των ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων στη Frontex. Θα ήθελα επίσης να ξέρω πώς θα είναι υποχρεωμένες οι χώρες να εξασφαλίσουν τους πόρους, το προσωπικό, την τεχνική, τις τεχνικές υποδομές. Ε, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον εισηγητή για αυτό το θέμα. Η κυρία Σπινέλη παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θεωρώ ότι προστατεύεται η Ευρώπη από αυτή την ε, συνοριοφυλακή η οποία είναι ένας μηχανισμός απέλασης. Είναι παράξενο που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτές τις λέξεις εδώ στην Ευρώπη. Και ότι αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να ε, συμπεριλαμβάνει στοιχεία όπω είναι η δικαιοσύνη όταν κάνουμε λόγο για ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί και οι θεμελιώδη δικαιώματα, γιατί και οι μπορούν να πετύχουν ε, αποτελέσματα και να είναι αποτελεσματικέ. Ευχαριστώ λοιπόν όλου για την παρουσίαση και τον εισηγητή και τον κύριο Λετζέρη. Ευχαριστώ. Διότι είναι πράγματα τα οποία με προβληματίζουν όλους ιδιαίτερως αυτά που αναφέρθηκαν όσον αφορά την πρόταση για την επικαιροποιημένη φρόντεξ αν θέλετε, και τον έρχο των συνόρων. Το περιθώριο, περιθώριο λιγμών και αρμοδιότητες μου προβληματίζει. Το περιθώριο λοιπόν κινήσεων των ομάδων παρέμβασης είναι κάτι που με προβληματίζει. Μπορούν να παρεμβαίνουν στις χώρες για επαναπατρισμό και χωρίς την συμφωνία των ελόγω κρατών μελών και αν τα κράτη-μέλη και αν συγκεκριμένα κράτη-μέλη είναι αντίθετα με αυτή την προσέγγιση. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει ακριβώς αυτό. Διότι αντιμετωπίζουμε ένα άλμα ομοσπονδιακό αν θέλετε, όπως είπε ο συνάδελφος της Άλντε, όμως υπάρχουν ομοσπονδιακά άλματα που στην πραγματικότητα είναι άλματα αντιδημοκρατικά και κεντρικού χαρακτήρα που δεν έχουν καμία σχέση με τον ομοσπονδιακό χαρακτήρα. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι ομοσπονδιακό άλμα με την κλασική έννοια του όρου. Το δεύτερο ερώτημα είναι οι αρμοδιότητες. Εδώ αναμειγνύονται η καταπολέμηση της τρομοκρατίας με την πολιτική ασύλου και με έναν τρόπο ακατανόητο για μένα όταν ο κύριος Λετζέρη αναφέρεται συγχώνευση μεταξύ του πυλώνα 1 και 2, θα ήθελα να γνωρίζω τι σημαίνει αυτό. Ε, χωρίς να υπάρχει καμία ρήτρα διαφύλαξη στη στιγμή που ένας οργανισμός, ένας φορέας, με έναν μόνο υπάλληλο που ασχολείται με τους μηχανισμούς καταγγελίας και προσφυγής σε περίπτωση παραβιάσεως δικαιωμάτων, πώς αυτός ο οργανισμός μπορεί να τα καταφέρει πολιτική εσωτερική ασφάλεια και πολιτική εξωτερική. Πώ μπορεί να τα ασκήσει όλα αυτά. Διότι να έχουμε ομάδε παρέμβαση σε τρίτε χώρε κατά τη τρομοκρατία είναι εξωτερική πολιτική. Αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μπάρμπαρα. Μπίρκιτ Σίπελ. Τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ Προέδρε. Πολλά ήδη υπόθηκαν. Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνική λοιπόν. Εάν συμφωνούμε ότι τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών μας είναι ευρωπαϊκά σύνορα, τότε βέβαια όλοι έχουμε κάποια ευθύνη. Και τότε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία είναι καλή ιδέα. Συγκεκριμένα ποιο είναι ο στόχος του φορέα αυτού, δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Αν θέλουμε να έχουμε ευρωπαϊκό οργανισμό, χρειαζόμαστε περισσότερους κοινούς κανόνες. Χρειαζόμαστε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Η ΔΕΜΗ είναι ανέφικτο να κινηθούν σωστά αυτοί που εργάζονται στον οργανισμό. Θέλω να φερθώ σε τρει τομεί, πέραν αυτών που ήδη αναφέρθηκα από συναδέλφου. Συμφωνούμε ότι εντό του οργανισμού χρειάζονται διάφοροι εμπειρογνώμονε για γλώσσα, μετανάστευση, έγκλημα. Κάποιοι θα εργάζονται εντό του οργανισμού, κάποιοι θα εργάζονται στα κράτη-μέλη και θα στέλνονται από τα κράτη-μέλη σε διάφορα σύνορα για να αντιμετωπίζουν επιτόπιε καταστάσει. Μιλάμε για πρόσβαση σε βάση δεδομένων. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι εμπειρογνώμονε οποιαδήποτε στιγμή θα έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων εθνική ή ευρωπαϊκή για οποιοδήποτε σκοπό ανα πάσα στιγμή. Τι είδου πρόσβαση εννοούμε, πλήρη πρόσβαση δεν καταλαβαίνω ποια θα είναι η διαδικασία. Έχω και ανησυχίες όσον αφορά τις εξουσίες του οργανισμού που δεν θα ισχύουν όλοι οι κοινοί κανόνες και ο διευθυντής τι εξουσίες θα έχει. Με ανησυχεί. Λείπει ο δημοκρατικός έλεγχος. Αυτό με ανησυχεί. Τρίτον. Δεν είναι θέμα αν μπορούμε να αποφασίσουμε γρήγορα ή όχι. Γιατί αξίζει να έχουμε γρήγορη απόφαση αν η υλοποίηση στην πράξη της αποφάσεως από τα κράτη-μέλη δεν γίνεται, αν λείπει. Πώς μπορούμε να πιστέψουμε ότι στέλνοντας μέλη προσωπικού από μια χώρα σε μια άλλη χώρα θα δώσει αποτελέσματα, αν τώρα βλέπουμε ότι πολλά κράτη-μέλη δεν στέλνουν προσωπικό στην Ελλάδα να εξασφαλιστεί η ταυτοποίηση και η καταχώρηση. Όλοι λέμε ότι είναι σημαντικό να κατοχωρηθούν όλοι αυτοί που έρχονται, να ταυτοποιηθούν, να ξέρουμε ποιο έρχεται. Τα κράτη-μέλη όμω δεν είναι έτοιμα να υποστηρίξουν αυτή την προσέγγιση. Πώ μπορούμε λοιπόν να πιστέψουμε, ακόμα και αν θεσπίσουμε αυτή την νομοθεσία, ότι τελικά στην πράξη θα λειτουργήσει. Πολλά εκκρεμή ζητήματα υπάρχουν και ερωτηματικά. Εγώ τι θέλω, αν δημιουργήσουμε μια νέα υπηρεσία, θα πρέπει να επικεντρωθούμε επί καλής νομοθεσίας, όχι γρήγορης νομοθεσίας. Και τέλος πρέπει να δούμε ποιος πληρώνει για όλες τις προσπάθειες. Το να στέλνουμε κόσμο από το ένα μέρος στο άλλο. Όλα πληρώνονται από τον παρόντα ευρωπαϊκό προπολογισμό. Τότε διαρωτώ με αν ισχύει κάτι τέτοιο. Ποιο ποσό θα παραμείνει για τους άλλους τομείς που χρειάζεται χρήματα από τον προπολογισμό. Πολλές ερωτήσεις ακόμα παραμένουν ε, αναπάντητες. Καλώς, λέει ο Πρόεδρος, να προσπαθήσω να συνοψίσω. Ε, ξεκινώ από εκεί που σταμάτησε η κυρία Σίπελ. Οι δημοσιονομικές συνέπειες αυτού είναι τεράστιες. Δεν θέλω να απολογούμε για το γεγονός ότι μέλη και οι παρουσιάζουν λεπτομερέστατα τις θέσεις τους, τις θέσεις της ομάδας και τι προσωπικέ τους. Τροφοδοτούν καλά τον εισηγητή και άρχισε τον κόπο η κουβέντα. Παρόλο που κράτησε πολύ η συζήτηση. Που δεν ήθιστε Δευτέρα βράδυ στο Στασβούργο, ξέρω ότι ο κόσμο είναι κουρασμένο, Άξιζε όμως τον κόπο να το κάνουμε. Διότι νομοθετικά δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια χρονικά για το θέμα. Θα ζητήσω από τον εισηγητή να ανακάμψει. Συνάδελφοι, έχουμε την αίθουσα μέχρι 21 και 30. Δεν θέλω όμως να μιλάει μόνο σε μένα κυρία Βουτσαμ και κανένας άλλος να είναι παρόν. Λοιπόν, παρακαλώ κάπως να μαζευτούμε χρονικά. Να πιστέψω στον κύριο Πάπριξ. Α, πριν από αυτό, θέλω να με κατευθύνετε κάπως. Είχαμε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Κάποιες ήταν ρητορικά σχήματα, θα έλεγα. Ρητορικά ερωτήματα, απευθυνόμαστε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, και κάποια πιο συγκεκριμένα από το ΤΠΕΣ Αλλά δεν μπορούμε τώρα να ακούσουμε εκτενείς ε, ομιλίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε, μπορείτε να απαντήσετε εν συντομία από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εν συντομία. Ποιος αλλούς ήταν? Ο κύριος Λετζέρη που άκουσε υπομονετικά σα όσα ελέγχθησαν και μετά θα επιστρέψουμε στον εισηγητή, αν συμφωνείτε. Εντάξει, κύριε Πάπριξ. Πρώτα ο κύριο Ντεκόιστερ, μετά ο κύριο Λετζέρι και μετά θα επιστρέψουμε στον κύριο Πάπριξ. Και παρακαλώ να μείνετε, συνάδελφοι, μην φύγετε για να μπορέσουμε να ακούσουμε. Να ακούσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομο. Δεν είμαι σίγουρο αν κατάλαβα όλε τι ερωτήσει και ποια είναι η φύση του, αν είναι ρητορικέ ερωτήσει ή πραγματικέ ερωτήσει. Τι εννοώ ρητορικέ ερωτήσει ότι θα υποβληθούν ερωτήσεις βάσει των όσων είπε το μέλος θέτοντα αυτά τα θέματα. Απαντήστε ό,τι θεωρείτε ότι μπορείτε να απαντήσετε εντό διλέπτου ή τριλέπτου. Θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω να διατρέξω τις ερωτήσεις δίνοντας κάποιες εξηγήσεις. Κοινή ευθύνη. Και μήπως κάποιες ευθύνες δεν είναι σαφείς και κάποια στοιχεία παραμένουν ακάλυπτα βάσει ευθυνών. Όταν μιλάμε για κοινή ευθύνη, πρώτη στη ευθύνη για τη διαχείριση εξωτερικών συνόρων ε, ανήκει στα κράτη-μέλη. Και τα καθήκοντα και αρμοδιότητε του οργανισμού παρατίθενται εξαντλητικά στην πρόταση. Άρα πρέπει να είναι πάντα σαφέ ποιο είναι υπεύθυνο γιατί. Σχετικά με ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία αυτών, δεν υπάρχει κενό. Πάντα πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Εάν δεν σαφέ το κείμενο του άρθρου 7, να το εξετάσουμε. Αλλά υπάρχει σαφή έρευνα και διάσωση. Αυτή η έκφραση χρησιμοποιήθηκε από αρκετού ομιλητέ. Η έρευνα και διάσωση. Από την περιγραφή του καθήκοντος που ανατίθεται στον οργανισμό στο άρθρο 7 αναφερόμεθα σαφώς σε κατεπίγουσες ανάγκες ανθρωπιστικής φύσεως και έρευνα και διάσωση που αποτελεί κομμάτι δράσεω που δρομολογείται από τον οργανισμό. Σχετικά με αυτό, ο κ. Κοέλιο μίλησε. Αναφέρθηκε στον κανονισμό του 2014 για τον νόμο των θαλασσών κάτι που αναφέρεται στο άρθρο 15 για το υπηρεσιακό σχέδιο. Δεν το λησμονήσαμε. Τα κάτι μελη υπέχουν την υποχρέωση να σεβαστούν τον κανονισμό και οργανισμό το ίδιο όταν ετοιμάζουν επιχειρησιακό σχέδιο. Αρκετοί αναφέρθηκαν στο εξή. Τι γίνεται αν χρειάζεται κατεπίγουσα δράση. Σύμφωνα το άρθρο 18, όταν το κράτο μέλο δεν συνεργάζεται, πρέπει να είμαστε σαφέστατοι. Ίσως να κρύβεται κάπως το κείμενο, το νόημα. Οι Frontex ή ο νέο οργανισμό δεν θα μπορούν να στείλουν τα στατεύματά του αν το κράτο μέλο το εν λόγω δεν συνεργάζεται όσον αφορά το επιχειρησιακό σχέδιο και δίνοντας οδηγίες και δίνοντας εντολές στους ε, αρμοδίους. Τα κυρίαρχα δικαιώματα του κράτους γίνονται σεβαστά. Με τα χαρά είδαμε ότι και ο εισηγητή και στο Συμβούλιο όμως κινούμεθα προ την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, στο άρθρο 26 του μηχανισμού Σέγγεν για τα σύνορα, αν το κράτο μέλο που χρειάζεται να δράσει ή χρειάζεται βοήθεια, δεν δράσει ή δεν ζητήσει βοήθεια, τότε πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προτείνει προς το Συμβούλιο επανεισαγωγή εσωτερικών ελέγχων συνόρων. Για τον προπολογισμό, εντέθησαν κάποιε ερωτήσει. Να επενθυμίσω το σημαντικότερο στοιχείο. 2016, επιδότηση για τη Frontex. 238 εκατομμύρια εγκρίθηκαν. Λάβαμε υπόψη την αύξηση που χρειάστηκε το 2015, τριπλασιασμός του προπολογισμού του Ποσειδών και του Τρίτων για να σώσουμε περισσότερες ε, ζωές εκείνων που κινδυνούν στη θάλασσα. Βασιστήκαμε σε αυτό. Το 2020 θα έχουμε 322 εκατομμύρια. Αύξηση. Δεν δεν τη θεωρώ και τόσο τεράστια αύξηση σε σχέση με το υψηλό επίπεδο που έχουμε σήμερα. Για στελέχωση αύξηση από 400 σε χίλιους ανθρώπους σταδιακά τα επόμενα χρόνια ούτω ώστε ο οργανισμός να μπορεί να απορροφήσει το νέο προσωπικό. Για το προπολογισμό αναφέρθηκε η ιδέα ξεχωριστών κονδυλίων. Εγώ για τα θέματα προπολογισμού δεν είμαι ειδικό. Η οικονομική αυτονομία του οργανισμού ίσως να επηρεάζεται. Χρειάζεται ε, λεπτομερής εξέταση. Κανονικά είναι ένα κονδύλι που εγκρίνεται για το οργανισμό και ο έλεγχος από το Κοινοβούλιο είναι εφικτός βάσει του, ε, του εγγράφου ενιαίου προγραμματισμού που έχει πολυετή συνιστόσα και αιτήσια συνιστόσα και μέσω της εκθέσεως δραστηριοτήτων που υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο. Ετέθησαν και πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Αφορούσαν το άρθρο 26. Μια ερώτηση. Πληροφορίες που μπορεί να δώσει ο οργανισμός στα κράτη-μέλη σε περίπτωση επιστροφών. Αυτή η διάταξη για μας είναι μια γενική αναφορά σε πληροφορίες. Είναι γενικόλογη. Μπορεί να αφορά και τι αρχέ τι οποίε απευθυνόμαστε σε τη χώρα για την απόκτηση ταξιδιωτικών εγγράφων κλπ. Ένα παράδειγμα. Και τα hot spots. Η περιοχή του hot spot, hot spot area. Και ο συγγητή το ανέφερε και στο Συμβούλιο. Έχουμε την πολιτική έννοια του hot spot, του σημείου υποδοχή. Χρειάζεται σαφή ορισμό στο κείμενο και στην έκθεση του κυρίου Πάπριξ και στη συμβαστική λύση του Συμβουλίου υπάρχει ένα ορισμό Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι από αυτού. Όταν ένα κράτο μέλο αντιμετωπίζει τόσο υψηλέ πιέσει στα εξωτερικά σύνορα, τα hot spots, η προσέγγιση των hot spots μπορεί να ακολουθηθεί. Αλλά hot spot, με την αυστηρή έννοια του όρου, μπορεί να είναι κάπου αλλού. Από εκεί που καταφθάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αν αποβιβάζονται σε κάποιο λιμάνι οι άνθρωποι, ο τόπος καταχωρήσεως και το κέντρο υποδοχής και γίνεται ο έλεγχος υγειονομικό, όπου γίνεται η ταυτοποίηση και τα δαχτυλικά αποτυπώματα μπορεί να είναι σε άλλη τοποθεσία. Αυτό φορά τον ορισμό που θα πρέπει να συμφωνήσουν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, δηλαδή πώς αυτή η έννοια θα ερμηνευθεί σωστά και θα διδυπωθεί ξεκάθαρα σε νομοθετικό κείμενο. Μου ζητήσατε να είμαι λακωνικός Πρόεδρε. Ελπίζω ότι απάντησα σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Απάντησα. Συγγνώμη που σας συντομεύω. Τώρα αποχωρούν τα μέλη και θα ήθελα να έχει κάποιο να τον ακούνε ο κ. Πάπρεξ. Ελπίζω, λέει ο να μην φταίει να μην φταίνει η απαντήση που φεύγει ο κόσμο. Ω, θα μπορούσατε να απαντήσετε πολλέ ερωτήσει ακόμα, ε, λέει ο πρόεδρο. Κύριε Ρετζέρη, θα πάτε αύριο σε συνεδρίαση των σκιωδών. Ευχαριστώ που ακούσατε τα μέλη. Μπορείτε να απαντήσετε κάποιε συγκεκριμένε ερωτήσει που σα απευθύνθησαν ε, εν συντομία, αν θέλετε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να απαντήσω στις ερωτήσεις που ετέθησαν όσον αφορά το ρόλο του οργανισμού για την ε, προστασία των εξωτερικών συνόρων. Ο ρόλος του οργανισμού της Frontex σήμερα δεν είναι μόνο να ελέγχει τον, τη μετανάστευση κυρίως την παράτυπη, αλλά έχει και έναν άλλο ρόλο που είναι καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και όλο και περισσότερο καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Θα σας δώσω κάποια πρόσφατα παραδείγματα όπου αναπτύχθηκε η υπηρεσία μας. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε ένα πιο σαφές νομικό πλαίσιο για παράδειγμα, όσον αφορά την εφαρμογή των ε, κοινών δικτών κινδύνου. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις πέρυσι, το Συμβούλιο ζήτησε η Επιτροπή και η Europol να αναπτύξουν κοινούς δείκτες κινδύνου προκειμένου να εντοπίζουν τους ε, ξένους μαχητές. Δεν μιλάμε για υπηκόους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάνε σε χώρες όπου μαθαίνουν να πολεμάνε, να γίνουν τρομοκράτες και μετά επιστρέφουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Frontex λοιπόν κλήθηκε να συνεισφέρει στον εντοπισμό τους. Αναπτύξαμε λοιπόν κάποια προγράμματα κι εμείς για να διαδώσουμε τις βέλτιστες πρακτικές προκειμένου στα διάφορα περάσματα συνόρων, εδώ δεν μιλάω μόνο για τα hot spots ή για τους παράτυπους μοτανάστες, αλλά για τα σύνορα, εκεί από όπου νόμιμα οι ταξιδιώτες περνάνε από τη μία χώρα στην άλλη, είτε διαξηράς είτε διαθαλάσσεις. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Αναπτύξαμε όμως και συνεργασία με το Europol και έτσι η υπόθεση στο μέλλον ότι αν έχουμε ένα χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας, το εξωτερικό σύνορο μπορεί ή πρέπει να χρησιμοποιείται ως φίλτρο όπου να εντοπίζονται οι ενδυνάμει απειλές και εδώ δεν μιλάμε μόνο για ξένους ή για μετανάστες αλλά μιλάμε και για Ευρωπαίους πολίτες. Αν καταζητείτε κάποιος Ευρωπαίος πολίτης από το δικαιοσύνη, από την αστυνομία σε μια χώρα μέλος είναι κρίμα να μην μπορούμε να το σταματήσουμε όταν αυτός βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή αυτή. Η Frontex λοιπόν έχει ως στόχο να στηρίζει τα κράτη-μέλη στα εξωτερικά σύνορα, στα σύνορα ή στα hot spots. Ο ρόλος του οργανισμού λοιπόν είναι να συνεργάζεται με τις αρχές επιβολής του νόμου, είτε πρόκειται για τα τελωνία, είτε για την αστυνομία, και να δίνει πληροφορίες και στοιχεία στη Europol και τη Eurojust. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε και εμείς να προχωρήσουμε όπου να μην υπάρχει πια πρώτος ή τρίτος πυλώνας, αλλά ο στόχος για καλή λειτουργία των εξωτερικών συνόρων. Όσον αφορά την πολιτική επιστροφών, εδώ να επιβεβαιώσω αυτό που είπε είπε και ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ρόλος της Frontex και στο μέλλον του νέου αυτού οργανισμού, συνοριοφυλακής και εκτοφυλακής, είναι να βοηθάει τις χώρες μέλη στην εφαρμογή των συμφωνιών ε, εισδοχής με μη ευρωπαϊκές χώρες. Ο ρόλος της υπηρεσίας μας είναι πολύ σημαντικός. Αν οι μετανάστες ε, καταγράφονται, ταυτοποιούνται στα hotspots και μετά αν τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται άμα τη στα hotspots μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αυτό μπορεί να βοηθήσει και ε, για τον σκοπό επιστροφής τους, αν τελικά αυτή προκύψει. Άρα λοιπόν ο μηχανισμός αυτός μπορεί να βοηθήσει τις ε, χώρες μέλη να έχουν ένα πασέλεσαι από τρίτες χώρες. Πρόεδρο, Διακόπτη, αύριο θα πάτε στη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών, σωστά, και εκεί θα συμμετάσχετε. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Επειδή δεν έχουμε χρόνο, θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Πάμπριξ, όσο έχουμε ακόμα εδώ τον κόσμο. Κύριε Πάμπριξ, εσείς. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ όλους σας για τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Οι περισσότερες ερωτήσεις ήδη απαντήθηκαν από την Επιτροπή. Πολλές από τις ερωτήσεις σας συζητήθηκαν σε βάθος μεταξύ των σχεδόν εισηγητών και όλων όσων συμμετείχαν στις συναντήσεις μας. Άρα λοιπόν απαντήσεις υπάρχουν στις περισσότερες από τις ερωτήσεις που ακούστηκαν. Η δουλειά συνεχίζεται και θα ήταν αφελές να πούμε σήμερα ότι το εγκρίνουμε, το ψηφίζουμε σήμερα. Όχι, θα συνεχιστεί η δουλειά. Και ό,τι καλές προτάσεις υπάρχουν θα συζητηθούν σε βάθος μεταξύ των σχεδόν εισηγητών. Κάποια σημεία όμως που θέλω να υπενθυμίσω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσει. Πρώτον, πρέπει να καταλάβουμε, όπω είπα και στην αρχή, ότι δεν πρόκειται για το φάρμακο που γιατρεύει τα πάντα, δεν είναι πανάκια. Δεν πρόκειται να λύσουμε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα με τη δημιουργία του νέου οργανισμού. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα βήμα μόνο. Και αν κάνουμε αυτό το βήμα και πετύχει, θα μπορέσουμε να κάνουμε και το επόμενο. Επίσης, θέλω να πω στην κυρία Σίπελ ότι Εάν εγκρίνουμε το κανονισμό αυτό, θα τεθεί σε εφαρμογή, θα φροντίσουμε γι' αυτό. Το πιστεύω. Και λέω, ναι, χρειαζόμαστε συμβιβασμούς στο Κοινοβούλιο. Γιατί το Κοινοβούλιο μας αποτελείται από διαφορετικές πολιτικές ομάδες. Το βλέπουμε. Κάποιες θα θέλαν επιστροφή στα εθνικά σύνορα. Κάποιοι άλλοι ακολουθούν το Imagine του Τζον Λένον και δεν θέλουν καθόλου σύνορα. Πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα σεβασμό που να είναι αποτελεσματικός, που να λειτουργεί, αλλά πρέπει να το κάνουμε και σύντομα. Γιατί η καθυστέρηση και η απουσία αποφάσεων δεν οδηγεί σε καλό αποτέλεσμα. Όσον αφορά άλλα θέματα, θα επανέλθουμε μεταξύ των σχεδόν εισηγητών. Και πιστεύω ότι μαζί θα βελτιώσουμε το κείμενο μέσα στους επόμενους μήνες. Και οι περισσότεροι από εμάς θα είμαστε ικανοποιημένοι. Κάποιοι και η κυρία Λάρουστιν ρώτησε κάποια πράγματα. Ευχαρίστως διμερώς να σας απαντήσω. Είναι σύντομη η προθέσμη για τροπολογίες. Είναι 20 Απριλίου στις 2 ώρα το μεσημέρι. Να ευχαριστήσω και τους και ηγητές και τους ε, ευρωβουλευτές που α, παρέστησαν εδώ και που συνεργάστηκαν και τώρα θα επανέλθω στο τελικό σημείο της Μεσσίας διάταξης που είναι είναι ε, έχει να κάνει με τι προποθέσει εισόδου και διαμονή υπηκών τριτών χωρών με σκοπό την έρευνα, τη σπουδέ, την ανταλλαγή με αυτών, την έμιστη και την άμιστη πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία και την απασχόληση των εσωτερικών άμιστων βοηθών. Ο λόγο στην Σεσιλία Βίξτρομ. Είσαι έτοιμη, Σεσιλία. Έχει ακόμα ενέργεια. Δεν θα γίνει κάποια παρουσίαση. 20 Απριλίου είναι η προθεσμία. Ευχαριστώ, Κλοντ, αγαπητοί συνάδελφοι, καθώς κάποιοι φεύγετε. Ελπίζω ότι αυτοί που σας απασχολεί το θέμα θα παραμένετε μερικά ακόμα λεπτά. Έχουμε καιρό συζητήσουμε για το θέμα των φοιτητών και των ερευνητών και τόσο στα όσο και εγώ έχουμε μεταβεί σε άλλα θέματα πετύχαμε μεγάλη πλειοψηφία πριν από μερικού μήνε στον Τρίλογο, όμω θα ήθελα και σήμερα να δράξω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω την ε, Προεδρία του Λουξεμβούργου, την Επιτροπή και προπάντων του σκιώδη συζητητή και ολόκληρη εβδομάδα μετά την πολιτική συμφωνία. Ε, ολοκληρώθηκε το κείμενο και το Συμβούλιο ανέκρινε ε, το σχέδιο. Επομένω, ε, οδεύουμε προς ε, την ψήφιση 1η ε, Μαΐου στην Ολομέλεια. Πρέπει να σας πω ότι τίποτα ουσιαστικό δεν έχει αλλάξει κατά τη διάρκεια αυτής της τελειοποίησης, του καθαρίσματος του κειμένου, των λέξεων, των κομμάτων κλπ έχουμε το ίδιο πολιτικό αποτέλεσμα στο κείμενο όπως και μετά την ολοκλήρωση του τριλόγου. Αυτό είναι βέβαιο. Είναι αυτονόητο. Υπάρχει όμως ένα ακόμα τεχνικό βήμα που ακολουθούμε για την πρώιμη δεύτερη ανάγνωση. Αν και θέλουμε ότι είμαστε σχεδόν έτοιμοι, θα Ελπίζω ότι όλοι θα υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία ώστε να προσελκύσουμε τους πιο ευφύς φοιτητές και ερευνητέ ώστε να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Θεωρώ ότι πετύχαμε καλούς συμβασμούς που απλοποιούν ε, τις διαδικασίες και αφαιρούν την γραφειοκρατία για πολλούς ε, ερευνητές και φοιτητές που θέλουν να έρθουν σε αυτή την Ήπειρο και να συνεισφέρουν. Ταυτόχρονα, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, δίνεται το εργαλείο στα κρατημέλη να αποφύγουν ε, ενδεχόμενες καταχρήσεις του συστήματος. Το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία είναι ευρύτερο και περιλαμβάνει όλους α, τους α, ειδικευόμενους, τους εθελοντές. Η κινητικότητα θα αυξηθεί και θα απλοποιηθεί και για φοιτητέ και για μέλη οικογένεια και για ερευνητέ και για ερευνητές και για μέλη τη οικογένειά του. έχουν και αυτοί το δικαίωμα να εργαστούν και επίση και οι φοιτητέ θα έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασία. Τώρα εισάγουμε ένα σύστημα που θα δώσει την ευκαιρία στου φοιτητέ και στου ερευνητέ να μείνουν τουλάχιστον 9 μήνε νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ολοκλήρωση των σποδών του ώστε να μπορέσουν να βρουν εργασία ή να ξεκινήσουν κάποια επιχείρηση και θα κάνουν πλήρη χρήση δυνατότητα και εμεί θα κάνουμε πλήρη χρήση φυσικά του δυναμικού αυτών των έξοχων μυαλών. Είναι η πρώτη φορά που αναφέρονται και οι όπερ, οι άμυστες βοηθοί. Είναι η πρώτη φορά που αναφέρονται και που τους παρέχεται κάποιο είδους προστασία. θεωρούμε ότι είναι πολύ βασικό ε, να διασφαλίζουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων. Και καθώς τώρα εστιάζουμε στην πολιτική ασύλου για προφανείς λόγους, είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε νομοθεσίες που θα αφορούν τις νόμιμες οδούς μετανάτευσης. Σας ευχαριστώ και καθώς ήδη έχουμε καθυστερήσει και το έχουμε συζητήσει το θέμα ε, και στο παρελθόν ε, αναμένω να υπάρξει μια θετική έκβαση της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Σεσίλια. Ανέφερα την προθεσμία για τους βουλευτές, για τους Είναι πολύ ευαίσθητο φάκελο όσον αφορά την νομοθεσία και αναφορικά με όλα αυτά που συμβαίνουν ε, αυτόν τον καιρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα 7, τους 7 ευρωβουλευτές που έμειναν στη θέση τους και παρακολούθησαν αυτό το τελευταίο σημείο της Ευρωπαϊκής ε, Ημερησίας Διάταξης. Να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε αυτό το τελευταίο σημείο. Θα ήθελα κάποιος να πάρει το λόγο. Δεν είμαι σίγουρος να θα το επιτρέψω. Όχι, δεν μπορώ να το επιτρέψω. Το έλαβα το μήνυμά σας. Θα θέλετε να πείτε κάτω. Θα είμαι σύντομη, γιατί προσπαθώ το ΕΛΚ, που είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Ε, καλωσορίζουμε αυτή την οδηγία και να εκφράσουμε την υποστήριξή μας την στην εισηγήτρια και να συμφωνήσουμε για την εξαιρετική δουλειά. Δεν θα θα πω απλώς γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο γιατί ε, αποσκοπεί στο να προσελκύσουμε και να κρατήσουμε ταλέντα που τα χρειαζόμαστε. Έχει να κάνει με την απασχόληση, ε, την αντικονιστικότητα, καθώς ε, η κοινωνία μας βασίζεται στη γνώση. Φυσικά θα υπάρξει και άρση της γραφειοκρατίας και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ καλό που οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να παραμείνουν στην Ευρώπη μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, γιατί αυτό έχει αποτελέσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, όπω καταλάβατε ήμουν πάρα πολύ σύντομη. Σα ευχαριστώ όλε. Τώρα μπορείτε όλες να είστε σύντομοι. Η κυρία Φαγιόν άνοιξε τη συζήτηση η Αναμαρία. Ευχαριστώ πολύ όλους και τη Σεσίλια και τους άλλους συναδέρφους. Ήταν σκληρό έργο, είναι ένα από τα σπάνια έγγραφα τα οποία επιτρέπουν με νόμιμους τρόπους να φέρουμε κόσμο στην Ευρώπη. Σεσίλια, ξέρω ότι κάνεις μια καταπληκτική δουλειά. Ήταν δύσκολο σεβασμός για όλους, αλλά έχουμε φτάσει σχεδόν στο τέλος. Ωραία, Τάνια, ευχαριστούμε. Μαρή Κριστίν Βεριζιά. Ναι, θα είμαι σύντομη, Πρόεδρε, το υπόσχομαι. Η ΓΚΟΕ συχνά είναι αυστηρή όσον αφορά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση. Εδώ όμως νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα προκειμένου να υπερψηφίσουμε το κείμενο και δεν πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Απλώς δεδομένου των υπόλοιπων πολιτικών της Ευρώπης για το μεταναστευτικό θα πρέπει να κάνουμε παραπάνω προσπάθεια για να προσελκύσουμε νέα ταλέντα. Η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι πολλοί νέοι από τις χώρες του Νότου φεύγουν να σπουδάσουν στην Αυστραλία, στον Καναδά, στις Ηνωμένε Πολιτείε, στην Τουρκία και δεν μένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ αυτό λοιπόν το βλέπω, το κείμενο δηλαδή, σαν μια πρόοδο απέναντι στις άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές. Πρόεδρος, ωραία, σωστά, τα λες, Να προσθέσω δύο άλλες διαστάσεις. αυτοί που επιστρέφουν στις χώρες τους πρέπει να βοηθιούνται για να χτίσουν τις χώρες τους και πάλι. Έχουμε 140 Σύριους φοιτητέ που τους έφερε ο πρόεδρος Σαμπάγιο στην Πορτογαλία. Φοιτητέ οι οποίοι εκτιμούν αυτό που τους προσφέρεται και θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους να την ανοικοδομήσουν. Άρα δεν είναι μόνο προς το δικό μας το συμφέρον, είναι και προς το συμφέρον των χωρών αυτών όταν θα υπάρξει εκεί η ειρήνη και πάλι. Και κάτι άλλο. Όπως είπε και η Τάνια, αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα είναι ότι δίνοντας προτεραιότητα στην ε, ανοποίηση των οικογενειών τους και αυτό θα πρέπει να είναι για μας προτεραιότητα. Είναι αυτό που ζητούν, αυτό που ζητούν οι οικογένειες των Σύριων ε, φοιτητών για παράδειγμα και θα πρέπει και αυτό να αντικατοπτρίζεται στο κείμενο της Σεσίλια. Πρόεδρος, ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ωραία, διάφορα. Τίποτα άλλο, επόμενη συνεδρίαση. Τρίτη, 12 Απριλίου, 11 και 4. Αύριο δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ όλους. Ευχαριστώ Σεσίλια.